Okay, friends. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση μας την απογευματινή. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον αντιπρόεδρό μας, τον Μάρος Σεφτσοβιτς. Εμείς τον προσκαλέσαμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πεδέχθη την πρόσκληση και είναι εδώ. Μας ενδιαφέρουν τα σχόλιά σας σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην Ενεργειακή Ένωση. Και φυσικά, μια και πρόκειται για Επιτροπή Απασχόλησης, μας ενδιαφέρουν και οι απόψεις ε, για τις συνέπειες που θα, έχουν, θα έχει στην απασχόληση η ενεργειακή μετάβαση και τι αντίκτυπο θα έχει στα ποσοστά ανεργίας αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Καλώς ήρθατε κυρία Αντιπρόεδρε. Μετά την εισαγωγή σας θα προβλέψουμε ένα χρόνο για συζήτηση με τους Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας, την πολύ ευγενική πρόσκληση, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε στο πρόγραμμά μας την οικονομική και κοινωνική διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης. Και θυμάμαι τι καρποφόρα και επικοδομητική συζήτηση είχαμε με τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Συμβούλιο. Και σας είμαι υπόχρεος που θέσετε και στο θέμα στην ημερήσια διάταξη και με προσκαλέσατε για συζήτηση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιουνκέρ, και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμένα διάλεξαν το σχέδιο της ε, Ενεργειακής Ένωσης ως βασική τους προτεραιότητα. Μέσω της Ενεργειακής Ένωσης ε, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από ένας απλός συντονισμός των ενεργειακών πολιτικών. Θέλουμε μια πιο σφαιρική, περιεκτική προσέγγιση πιο ολιστική όπως λέμε, γιατί όταν μιλούμε για την ενέργεια δεν είναι μόνο η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωσή της, αλλά πώς θα συνδυαστεί με τις άλλες μας πολιτικές η ενεργειακή πολιτική, πώς θα μειώσουμε τη, τα καυσαέρια, όχι μόνο από ε, την παραγωγή ενέργειας, αλλά και από τις μεταφορές, από τη γεωργία, πώς θα βελτιώσουμε, θα ενισχύσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων μας και δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας αν δεν είμαστε πιο προηγμένοι στην έρευνα, στην καινοτομία και αν δεν καταφέρουμε να θέσουμε στην εμπορία τις νέες τεχνολογίες. Δουλεύουμε λοιπόν ως ομάδα με πνεύμα συνεργασίας και θα σας παρουσιάσω τις τα αποτελέσματα της Ενεργειακής Ένωσης, τις εξελίξεις και τι επίπτωση θα έχει αυτή στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό θέμα προς επισήμανση είναι ότι γινόμαστε μάρτυρες της γνήσιας ενεργειακής μετάβασης εξαιτία των κλιματικών μας στόχων και εξαιτία των νέων τεχνολογιών που σας ανέφερα προηγουμένως. Επίσης είναι σαφές ότι αυτή η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει πρώτα απ' όλα φυσικά τον ενεργειακό τομέα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν. Για παράδειγμα, είμαστε μάρτυρες της μετάβασης σε μια οικονομία ε, ουδέτερη από άποψη άνθρακα. Δεν θα έλεγα απολαγμένη από άνθρακα, αλλά ουδέτερη από άποψη άνθρακα. Και στα πλαίσια αυτής της ενεργειακής μετάβασης επιδιώκουμε ένα πραγματικό εξυγχρονισμό της οικονομίας μας. Επίσης, σας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίε ε, για την επένδυση, για τις επενδύσεις, την απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση. Βέβαια προποθέτει αλλαγέ και προσαρμογή σε πολλού παραδοσιακού κλάδου τη οικονομία μα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και τι δύο πτυχέ, και τι ευκαιρίε, αλλά και τι προκλήσει. Και θα πρέπει να λάβουμε και τις δύο υπόψη. Θα ξεκινήσω με τις ευκαιρίες, αν μου επιτρέπετε. Το 2014 οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν μια αξιολόγηση του αριθμού των θέσεων απασχόληση που συνδέονται με τη μετάβαση σε ε, οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ήδη από το 2014 9 εκατομμύρια θέσει απασχόληση συνδέονταν με την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέχρι το 2030 η προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό στους τομείς αυτούς ε, θα είναι διπλάσιες. Δηλαδή θα μιλούμε για 18 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης από 9 που ήταν πριν στην Ευρώπη. Και αυτό αφορά ε, το θέμα της ζήτησης, όχι μόνο στα θέματα ενεργειακής απόδοσης, αλλά και στην, στις ε, τεχνολογίες για, την, για τη θέρμανση, για τον ηλεκτρισμό, με χαμηλή χρυσή άνθρακα, αλλά και στο θέμα της ενεργειακής αποθήκευσης, αποθήκευσης ενέργειας. Από το 2014 περνάμε σε μια νέα δυναμική και αυτό φάνηκε και από τη Συμφωνία των Παρισίων, μια συμφωνία που σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της παγκόσμιας κοινότητας να περάσει στη, σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι Οπότε, από τη μια θα γίνουν πολλές προσπάθειες για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μάλιστα τη στιγμή που οι παγκόσμιες ανάγκες ενέργειας θα αυξηθούν κατά 30% μέχρι το 2040. Αυτές είναι οι στατιστικές που προέρχονται από τον, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Φαίνονται αντιμαχόμενες και αντιφατικές αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά επειδή ακριβώς θα χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια, θα πρέπει η ενέργεια αυτή να προέρχεται από λύσεις και τεχνολογίες που δεν χρησιμοποιούν πολύ άνθρακα, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αυτό παγκοσμίω. Επίσης, στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α, το θέμα είναι τα κράτη-μέλη και οι βιομηχανίες μας θα δράξουν αυτή την ευκαιρία, είναι έτοιμες να την αξιοποιήσουν. Από αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό ε, η πορεία μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε και το ειδικευμένο προσωπικό. Το θέμα και οι προκλήσεις των δεξιοτήτων και των προσόντων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίω σε επίπεδο εκπαιδευτικών συστημάτων από τα κράτη-μέλη, σε επίπεδο βιομηχανία και κοινωνικών εταίρων. Αλλά ήδη μέχρι στιγμή ε, έχουν αναλυθεί αρκετέ πρωτοβουλίε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί και να ε, διαπιστώσουμε ότι αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται παντού, ούτε με την απαραίτητη ταχύτητα. Και εκεί ακριβώς πιστεύω ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα συμβάλλουν στο να ενταθεί η συζήτηση. Την περασμένη Παρασκευή οθετήσαμε το θεματολόγιο για τις δεξιότητες στην Ευρώπη. Αυτό το θεματολόγιο επικεντρώνεται σε οριζόντιες δεξιότητες και τη σημασία που έχει η πρόσβαση σε ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Χαίρομαι που η πρωτοβουλία αυτή συνδέει το θέμα των δεξιοτήτων με την Ενεργειακή Ένωση και τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Να σταθώ σε μερικά σημεία για αυτή την αλληλεπίδραση. Το θεματολόγιο των δεξιοτήτων προβλέπει ε, ε, μια πρωτοβουλία για διακλαδική συνεργασία για τις δεξιότητες. Έτσι θα κινητοποιηθούν και θα συντονιστούν βασικοί συντελεστές οικονομικών κλάδων, ώστε να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να χρησιμοποιηθεί με πιο στρατηγικό τρόπο ε, τα κοινοτικά κονδύλια και τα εθνικά κονδύλια. Και έξι τομείς έχουν επιλεγεί για πιλωτικά προγράμματα εξαιτία του βαθμού οριμασή τους. Ένας είναι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και ο δεύτερος είναι οι μεταφορές, οι τεχνολογίες, ε, οι θαλάσσιες τεχνολογίες και οι δύο αυτοί αναπτύσσουν όλο και πιο φιλοπεριβαλλοντικές και βιώσιμες τεχνολογίες. Ειδικά οι τεχνολογίες της θάλασσας περιλαμβάνουν και εγκαταστάσεις ε, αιωλικής ενέργειας και χρήσης της ενέργειας των κυμάτων και μάλιστα offshore. Βέβαια θέλουμε να επικεντρωθούμε και σε άλλους κλάδους με ε, επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πράσινη ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το μέσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, όπω είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτονόητο ότι είναι απαραίτητο. Επίση, ο οικοδομικό κλάδο, ο κατασκευαστικό κλάδο, θα πρέπει τα κτίρια που κατασκευάζουμε να είναι πιο ε, αποδοτικά από άποψη ενέργεια και να έχουμε και τι επιδομέ για πιο ε, αποτελεσματικές τεχνολογίες για τα, για τα δίκτυα διανομής, για την ε, θέρμανση της πόλης, ε, τηλεθέρμανση και ούτω καθεξής. Θέλουμε εφή κτίρια στις πόλεις μας και όλα αυτά πετούν νέες δεξιότητες για να συνδυάσουμε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και να τις προωθήσουμε από τη φάση της σύλληψης και του σχεδιασμού στη φάση της κατασκευής και της εμπορίας. Τρίτος τομέας που αναφέρθηκε ε, στο έγγραφο για το, για, τη θεματολογία των για το θεματολόγιο των ε, δεξιοτήτων. Η χαλιβουργία, ε, που είναι ένας κλάδος έντασης ενεργειακής, γι' αυτό και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο η τεχνολογία δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα για να μειώσουμε τις εκπομπές και επίσης συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και τις ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν των πρωτοβουλειών όμως αυτών που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειαζόμαστε αντίστοιχε και σε εθνικό επίπεδο. Ένα τμήμα της, στρα... της στρατηγικής μας για την Ενεργειακή Ένωση και των συναφών προτάσεων αφορούσε την προετοιμασία των εθνικών ενεργειακών και κλιματικών προγραμμάτων. Και αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως έγγραφα στρατηγικής που θα χρησιμοποιηθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις για να αναπτύξουν στρατηγική, για να διαχειριστούν την ενεργειακή μετάβαση και εγχώρια, να γίνει η διασύνδεση ε, και με τις θέσεις απασχόλησης και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίσης. Τώρα, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που χρησιμοποίησε η Κορίνα Κρέτσου η Επίτροπος πριν από μία εβδομάδα. Τώρα για το πώς ε, προσπαθούμε να στηρίξουμε μέτρα αποτελεσματικότητας, ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας στα κράτη-μέλη. Ήταν καλοπροαίρετο το πρόγραμμα, αλλά απέτυχε δυστυχώς και απέτυχε γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί ειδικευμένοι ε, εργαζόμενοι για να εγκαταστήσουν τις νέες τεχνολογίες. Οπότε, σε τελική ανάλυση, το πρόγραμμα χρειάστηκε να μετατραπεί σε πρόγραμμα που στηρίζει τη δημιουργία των δεξιοτήτων πρώτα για να περάσουμε στη συνέχεια στη δεύτερη φάση που είναι η χρήση αυτών των των εργαζομένων για να μπορούν να χρησιμοποιούν στην κατασκευή των κτηρίων τις νέες τεχνολογίες. Οπότε, ποιο είναι ο ρόλο των ενωσιακών κονδυλίων, τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση και το θεματολόγιο δεξιοτήτων και απασχόληση. Εμείς συμβάλλουμε ε, προκειμένου να δούμε και επί τόπου την ενεργειακή μετάβαση. Σημαντικά κονδύλια προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. 69 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά για την περίοδο 2014 μέχρι 2020 ε, που καλύπτει και τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης. Επίσης, ε, η πολιτική συνοχή ε, δεν περιορίζεται μόνο στα κονδύλια, στο οικονομικό σχέδιο, γιατί περιλαμβάνει και την εδαφική ανάπτυξη και ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει θέματα και τοπικά που αφορούν την ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, προσφέρουμε τεχνική αρρωγή για τη δημιουργία ικανοτήτων, ώστε οι επενδύσει αυτές να συμβάλλουν σε μια πραγματικά βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Πέρυσι είχαμε ε, βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές τεχνογνωσίας μεταξύ των κυβερνήσεων προκειμένου να ε, εφαρμόσουμε κάποια ενεργειακά προγράμματα που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει να δοθούν κάποιοι κονδύλια στην εκπαίδευση, στις υποδομές, ώστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να είναι συμπληρωματικό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γιατί τουλάχιστον 1,1 δις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα αφιερωθούν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για να γίνει η προσαρμογή των δεξιοτήτων που με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων κλάδων της ενέργειας και του περιβάλλοντος και των νέων αναγκών τους. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων μεταξύ των ερευνητών στα πλαίσια των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Πολλές χώρες και περιφέρειες δίνουν προτεραιότητα στην έρευνα τεχνολογική ανάπτυξη για στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα και έρευνα για την ενέργεια. Οπότε θέλουμε τέτοιε πλατφόρμε για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στι τελευταίε ε, ε, εξέλιξει και στι πιο σύγχρονε γνώσει. Ε, θέλουμε να βοηθήσουμε και τις περιοχές να προλάβουν και να διαχειριστούν τις συνέπειες της ενεργειακής μετάβασης. Αυτό ενδιαφέρει όλες τις περιφέρειες και κυρίως αυτές που εξαρτώνται ε, από ρηκτά καύσιμα. Κυρίως. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Ταμείο Juncker δηλαδή. Έχουμε ένα σχέδιο στον Καλέ για παράδειγμα, μια περιοχή που έχει παραδοσιακές βιομηχανίες και θέλουμε να συνδυάσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Ταμείο Juncker, και να χρησιμοποιήσουμε τη στήριξη αυτή, τη συνδυασμένη, για να αναπτύξουμε στην περιοχή μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα και χαμηλών εκπομπών και να μπορέσουν και οι περιφέρειες αυτές να αναπτύξουν οικονομίες με χαμηλή χρήση άνθρακα, με απότερο σκοπό να γίνουν περιφέρειες ε, με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Και ταυτόχρονα θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, να αναπτύξουμε γενικώ την οικονομία και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξελίξεις για να καταπολεμήσουμε την ε, αένδια των καυσίμων. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο ακόμη σχόλια που ευελπιστώ ότι θα τα αναλύσουμε πιο ενδελεχώς στην ακόλουθη συζήτηση. Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου είναι το πρώτο. Το 2015 είχα συναντήσεις με διακλαδικούς εταίρους για να συζητήσουμε αυτό το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης. Πολύ χρήσιμες αυτές οι δύο συναντήσεις και θα συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτούς τους διαλόγους υψηλού επίπεδου με κάποιες ε, τομεακές πρωτοβουλίες. Και αυτό το blueprint που σας ανέφερα θα ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους στους διαφόρους κλάδους να εγγύψουν σε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος το θέμα της ενεργειακής ένδυας, ενεργειακής παινίας. Το συζητήσαμε και στην Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες Εκεί φάνηκε η σημασία αυτού του θέματος και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όχι μόνο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε επισταμένως τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να τις ε, ενστερνιστούμε, τουλάχιστον στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Αυτά κυρία Πρόεδρε προς το παρόν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνω μια απόπειρα με σύντομη επισκόπηση των οικονομικών ευκαιριών και προκλήσεων που μας δίνει αυτό το σχέδιο της Ενεργειακής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στην κυρία Σαντέπρατα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχά, να σα πω ότι μιλώ εξ ονόματο του κ. Καζά, ο οποίο και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να προηγηθεί σήμερα το απόγευμα. Ο αριθμό λοιπόν των άνθρωπων που απειλούνται από ένδια και από κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη διαρκώ αυξάνεται. Και αυτή η ένδια προφανώ πάει χέρι-χέρι με μια επισφάλεια ενεργειακή. Το θέμα λοιπόν είναι πώ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Και νομίζω ότι καταρχάς λιγότερη ακριβή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Και η αποδοτικότητα ενεργειακή θα πρέπει να αποτελεί μία προτεραιότητα. Και η ΕΛΚ, το ΕΛΚ λοιπόν προτιμάει και προωθεί λύσει ε, προς την κατεύθυνση αυτή παρά ε, πιο πολύ κατασταλτικούς μηχανισμούς που θα ελέγχουν την κατανάλωση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, ιδιαίτερως αυτή των κτηρίων και πώς ε, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έξοδο από την επισφαλή κατάσταση για πολλά τέτοια νοικοκυριά. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα τιμολόγια τους, τους λογαριασμούς τους σε ό,τι αφορά την ενέργεια με βιώσιμες ε, ε, λύσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα και μόνο οικονομικές και θέλουμε να εισαγάγουμε και άλλα μέτρα και άλλα μέσα. Μεταξύ άλλων ε, μέτρα εκπαίδευσης των καταναλωτών τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση της πατάλης ενέργειας, αλλά και να βοηθήσουν τον καταναλωτή να ακολουθεί μια συμπεριφορά υπεύθυνη σε ό,τι αφορά και τα έξοδα και την ενεργειακή κατανάλωση. Έχετε ήδη απαντήσει κάποια από τα ερωτήματα τα οποία ήθελα να θέσω. Καταρχάς, ποιος ε, είναι ο ρόλος που μπορεί να διδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουν αυτά τα πρακτικά σημεία να εφαρμοστούν ε, σε ευρεία κλίμακα και κατά δεύτερον τι μέτρα θεωρεί ότι μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσει την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδυας. Μέτρα πέρα από αυτά που ήδη αναφέρατε. Μία άλλη ερώτηση, κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη φτώχεια μπορεί να που μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, αν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Τέλος, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερώσει, έχει επικροποιήσει τα δεδομένα προκειμένου να εντοπιστούν ποια άτομα ζουν σε αυτό το καθεστώς ενεργειακής επισφάλειας. Αυτό θα μας οδηγούσε σε καλύτερη και πιο στοχοθετημένη παροχή βοήθειας. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε προκειμένου αυτοί που απειλούνται να μπορέσουν να βοηθηθούν από μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής ε, ένδυας. Και φυσικά θα πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο και την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση. Η Γιούτα Στάινρουκ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Ξέρετε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το περίφημο κοινωνικό mainstreaming γιατί η απασχόληση και οι κοινωνικές επιπτώσεις ε, αυτά τα δύο είναι θέματα που ε, λαμβάνονται αλλού υπόψη πέρα από την πολιτική απασχόλησης. Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για την κυκλική οικονομία, για τις ε, πρώτες ύλες, το τι θα γίνει στο μέλλον και Αυτά όλα σίγουρα θα έχουν επιπτώσει στην πλήρη απασχόληση. Εσείς είπατε ότι προσδοκάτε ανάπτυξη και μέσα από την Ενεργειακή Ένωση. Μιλήσατε πολύ για τα συμφέροντα της οικονομίας. Εμείς έχουμε κατά νου και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ε, είπατε ότι θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξουν νέες θέσεις απασχόλησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτές θα είναι νέες, αλλά ότι υπάρχουν θέσεις απασχόλησης που αλλάζουν. Μερικές εξ αυτών εξαφανίζονται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να έχουμε ε, κατά το θέμα της απόκτησης δεξιοτήτων ε, στο σχολείο αλλά και στα πανεπιστήμια στην Ευρώπη δεν το καταφέρνουμε σε αυτό το θέμα τόσο καλά όσο σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αλλά η λέξη κλειδί είναι η διαβίου μάθηση. Διότι στις μεγάλες επιχειρήσεις, ε, εγώ έρχομαι από μια μεγάλη βιομηχανική πόλη με τη μεγαλύτερη χημική βιομηχανία στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να χρηματοδοτείται η διαβίου μάθηση στις επιχειρήσεις αυτές. Αλλά και στις μικρές, κυρίως στις μικρές, δεν υπάρχουν τέτοιες οικονομικές δυνατότητες δυνατότητες. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, η Κομισιόν έχει κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις απαραίτητες δεξιότητες. Μία άλλη ερώτηση. Εσείς ε, πώς ακριβώς προετοιμάζετε την αλλαγή των ε, θέσεων απασχόλησης. Πέρα από αυτά που μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Τάισεν σχετικά με το θεματολόγιο των δεξιοτήτων, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Όσον αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, χαίρομαι πάρα πολύ ε, που δίνετε σημασία στο θέμα αυτό. Εγώ έρχομαι από τη Γερμανία και στη τελική ανάλυση αυτοί είναι οι ειδικοί που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τους ε, πολιτικούς και την Κομισιόν τι ακριβώς και πώς πρέπει να διαμορφωθεί. Ε, δείξατε την ενεργειακή επάρκεια βλέπω ότι σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες υπάρχει ένα ε, ανεκμετάλλευτο δυναμικό για να προκύψει ανάπτυξη. Πριν από κάποια χρόνια εγώ ανακαίνισα το σπίτι μου με νέα ενεργειακά ε, πρότυπα και είδα πόσοι άνθρωποι απασχολήθηκαν ε, σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, εγώ ήμουν στην ευτυχή θέση να μπορώ να το χρηματοδοτήσω αυτό. Πολλοί όμως δεν μπορούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα δηλαδή το θέμα είναι ε, πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα επιτόπου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα στήξης. Το ίδιο ισχύει και για δήμους και κοινότητες ε, ε, που χρήζουν και έχουν ανάγκη από ανακαίνιση. Από την άλλη πλευρά όμως αυτές, ε, αυτοί οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν τόσα πολλά δάνεια που δεν μπορούν να επενδύσουν σε ανακαίνιση, βιώσιμη ανακαίνιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν όλοι σας οι συνάδελφοι. Οι πόροι αυτού σιγά σιγά εξαντλούνται. Νομίζω λοιπόν ότι τελικά όλοι οι τομείς ε, έχουν πολλές προσδοκίες ε, και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πάω στο θέμα της ε, ενεργειακής φτώχεια. Επ' αυτού θα μιλήσουν οι συνάδελφοι. Για μας όμως είναι σημαντικό οι θέσει εργασία που δημιουργούνται να είναι βιώσιμες, να είναι καλές. Και μόνο έτσι μπορεί να προκύψει ανάπτυξη και για τους πολίτες. You Ξεκινήστε αν θέλετε με τις απαντήσεις και θα συμπληρώσουμε τα ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα και να ευχαριστήσω και τους δύο βουλευτές για τις ερωτήσεις που έκανε η κυρία Σάντερ. Τόνισε τον ε, κίνδυνο ένδυας φτώχειας. Νομίζω ότι αυτό έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την πρόσφατη οικονομική κρίση και το γεγονός είναι ότι έχουμε κάνει αναλύσεις, αναχώρα και όλα αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σαφώς δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει πληχθεί από το πρόβλημα της ενεργειακής ένδυας. Αυτό πραγματικά έχει πληξει όλες τις χώρες και το γεγονός ότι υπάρχουν πάνω από 10% των Ευρωπαίων, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους που έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους, είναι νομίζω πολύ το στον 21ο αιώνα ότι αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα ενεργειακής ένδυας. Είναι λοιπόν αρκετά σαφές ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Και μάλιστα θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι εμπίπτει στο, στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι όταν ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα θέματα η ενεργειακή ένδια. Και αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε κατάρτιση εθνικών στρατηγικών, το τι θα πρέπει να κάνουν και τι προτίθεται να κάνουν τα κράτη-μέλη. Και πώς από το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να βοηθήσουμε με μια σοβαρή επικέντρωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί, όπως είπατε, πρόκειται για το πιο ασφαλή, πιο φθηνό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αν υπάρξει σωστή ενεργειακή αποδοτικότητα στα νοικοκυριά, στις μικρομισές και στις βιομηχανίες, θεωρώ ότι ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος και στα εργοστάσια θα υπάρχει δηλαδή πραγματικά εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος. Και ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για τις νέες ε, τεχνολογίες, είναι επιτετικές σε ό,τι αφορά την ένταση εργασίας. Θα θέλαμε λοιπόν αυτά να γίνουν από τις τοπικές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τους τοπικούς εργάτες και εργαζόμενους προκειμένου αφενός να αντιμετωπίσουμε δύο στοιχεία. Να σώσουμε τον πλανήτη, να εξοικονομήσουμε χρήμα για την ενέργεια που σπαταλάται και παράλληλα να δημιουργηθούν και θέσει εργασία για τι τοπικέ οικονομίε. Γιατί οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι αυτέ που θα εφαρμόσουν όλε αυτέ τι τεχνολογικέ συσκευέ για να υπάρχει ενεργειακή αποδοτικότητα. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε, Να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω να μην περιοριστούμε σε ενεργειακή αποδοτικότητα μιλώντα για τα κτίρια. Θεωρώ ότι πλέον έχουμε τι τεχνολογίε που μα επιτρέπουν να πετύχουμε ευφυή κτίρια. Κτίρια τα οποία θα εξυπηρετούν τον νέο σκοπό του 21ου αιώνα και τη σχετική οικονομία. Τέτοια κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αλλά και να αποθηκεύουν και να παράγουν ενέργεια που θα έχουν ηλεκτρικούς φορτιστές αυτοκινήτων, για παράδειγμα, κτίρια τα οποία θα μεταδίδουν σήμα σύρμα του ίντερνετ. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιες νέες πλατφόρμες, κτίρια για την ε, οικονομία των δεδομένων του 21ου αιώνα. Θα ήθελα να τονίσω ότι τον, ε, το φθινόπωρο θα υποβάλουμε ένα πακέτο για την ενεργειακή υποδοτικότητα και εκεί σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τη νέα ε, οδηγία για την ενέργεια αλλά και για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και θέλουμε αυτό να το συνδυάσουμε με την πρόταση για την ευφύ χρηματοδότηση ευφύων κτηρίων αλλά και με μια πιο στενή συνεργασία των ευφύων πόλεων με τις τοπικές αρχές. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για το θέμα της μίας και ενιαίας θηρίδας, one-stop shop για τις τοπικές αρχές. Δηλαδή, μέσα από μια ενιαία θηρίδα, μέσα από την ιστοσελίδα μας, θα, μπορούμε, θα μπορεί ο κόσμος να λαμβάνει συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει ζητήματα. Πώς να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, την οπική πτυχή και τις νομικές ε, περιπλοκές που συνδέονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έτσι θεωρώ ότι θα προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλη την Ευρώπη. Και αν θέλουμε να ωφεληθούμε από την οικονομική αυτή μεταμόρφωση θα πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση υψηλού επίπεδου, σε μια πιο καλή κατεύθυνση, αν θέλετε, των νέων. Ποια είναι τα επαγγέλματα, ποιες, ποια είναι τα προσόντα τα οποία θα χρειαστούμε στο μέλλον και τι προσόντα πρέπει να έχει κανείς για να βρει μια σωστή και βιώσιμη θέση απασχόληση στην αγορά. Νομίζω ότι αποκαινούμε τα κράτη-μέλη με τους ακαδημαϊκούς κύκλους και με τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να, αποφεύγουμε, να αποφύγουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, όπου εκατομμύρια νέοι πολύ συχνά με πολύ υψηλά προσόντα και πολύ υψηλή εκπαίδευση, απλά με προσόντα τα οποία δεν, δεν ζητούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία, μένουν άνεργοι. Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ατζέντα για τα νέα προσόντα για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν σωστές αναλύσεις και σωστές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Ποια θα πρέπει να είναι η γενική προσέγγιση, τι προσόντα χρειαζόμαστε. Πώς αυτό θα ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα και πώς θα δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες στους νέους. Σε ό,τι αφορά το σκέλος ε, της προστασίας του καταναλωτή και της ενεργειακής ένδυας. Ένας άλλος τομέας, τον οποίο θα πρέπει και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, ε, αυτό έχει να κάνει και με την ερώτηση που έκανε η κυρία Στάινρουκ. Είναι το εξή. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε και την πρόταση που θα δημοσιεύσουμε πριν τα τέλη του έτους για την ε, νέο σχεδιασμό του ρικρισμού όπου θα είναι πολύ πιο ενεργός ο ρόλος του καταναλωτή. Θα είναι σε θέση ότι ο καταναλωτής όχι μόνο να είναι καλύτερα ενημερωμένος, αλλά να καθορίζει και την ενεργειακή του μοίρα. Αν θέλει να καταναλώνει αλλά και να παράγει ενέργεια θα μπορεί να το κάνει. Αν θέλει να έχει πιο εύκολη πρόσβαση στις ανταγωνιστικές ενεργειακές εταιρείε να μπορεί να το κάνει. Εκδημοκρατισμός, λοιπόν, της ενεργειακής παραγωγής. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ πιο ενεργή προσέγγιση του καταναλωτή. Αυτό θα οδηγήσει, θεωρώ, σε πιο μεγάλο ανταγωνισμό και σε καλύτερα στη μέση του καταναλωτή. Ύστερα, τονίσατε το τι θα πρέπει να γίνει με τα προσόντα εκείνα, με τις θέσεις απασχόλησης εκείνες, οι οποίες συνδέονται με τις παραδοσιακές ε, μορφές παραγωγής και που εξαφανίζονται σιγά σιγά. Εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με ένα τέτοιο τρόπο, προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές τις οποίες τόνισα και στη συζήτησή μου με τους δημάρχους χθε, στην αντισυναντηθήκα με τους ε, δημάρχους των Ευρωπαϊκών Πόλεων θα πρέπει να σκεφτούμε εκ των προτέρων λίγο πώς θα τροποποιηθεί η κατάσταση και η θέση των πόλεων, των περιφερειών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παραδοσιακές ε, μορφές παραγωγής ενέργειας και να δώσουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο, μία εναλλακτική δυνατότητα με κάποια μορφή εκπαίδευσης, μεταεκπαίδευσης ενδεχομένως ή μέσω της διαβίου εκμάθησης να δώσουμε δεύτερες ευκαιρίες επαγγελματικές σε όσους θέλουν να αποκτήσουν νέα προσόντα, ιδιαίτερα από τα επαγγέλματα αυτά και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τονίσατε τη σημασία των τοπικών αρχών, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί αυτές είναι πιο κοντά στον πολίτη. Άρα, καταρτίζουμε νέα πλαίσια για βάση και τη αρχή των αθλίων πόλεων και βάσει και του συμφώνου του Άμστερνταμ που συμφωνήθηκε και έτσι ξεπεράστηκαν κάποιοι δισταχμοί που υπήρχαν μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ευρωπαϊκών πόλεων για να τονιστεί και η αρχή της επικουρικότητας και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, bottom up. Φυσικά χρειάζεται συνεργασία αλλά χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για να ανταλλάσσονται οι βέλτιστες τακτικές και να υπάρχει μια σωστή συνεργασία. Αυτή την πλατφόρμα λοιπόν θα προτείνουμε. Τελευταίο, χρηματοδότηση. Περιορισμένη είναι ασφαλώς παντού η δημόσια προπολογισμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, ξέρετε τι γίνεται και στα κράτη-μέλη άλλωστε. Τι ήθελα να τονίσω. Έκανα και πολλές συναντήσεις με τα συνταξιδοτικά ταμεία, με τους εκπροσώπους του χρηματοοικονομικού κόσμου, με τις πράσινες επενδύσεις, τον πράσινο κόσμο, όπως τον αποκαλώ. Μα λένε ότι, κοιτάξτε, εμεί έχουμε 3 εκατομμύρια να επενδύσουμε σε πράσινα προγράμματα. Δεν περιοριζόμαστε όπω οι τράπεζες, από τα ποσοστά απόδοση από την απόδοση του επόμενου έτος, αλλά χρειαζόμαστε μια σταθερότητα, χρειαζόμαστε μια στρατηγική πορεία και κατεύθυνση τη οικονομία και χρειαζόμαστε ασφαλώ και καλά έργα και ασφαλώς ε, μοιρασμένο κίνδυνο με κάποιον. Και νομίζω ότι έτσι προχωράμε με σωστό τρόπο με την Τράπεζα Επενδύσεων και νομίζω ότι αν πετύχουμε το μηχανισμό αυτό θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε πάνω από 100 δις σε ένα χρόνο και θα πρέπει όλες αυτές λοιπόν οι τέχνικες να χρησιμοποιηθούν για να μπορούν να αφιερωθούν όλα αυτά στις ευφύλες τεχνολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν τώρα Προηγουμένως όμως να σας δώσω μία πληροφορία γιατί διεξάγεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Σλοβακίας. Γι' αυτό είμαι τόσο νευρικός όπως βλέπετε, δεν μπορώ να καθίσω στη θέση μου. Ε, ένα μηδέν ε, προηγείται η Σλοβακία προς το παρόν πάντως. Ηρεμήστε. Οπότε τώρα έχετε και ανανεωμένη ενέργεια και φόρα. Το ίδιο και ο κύριος Κούκαν. Και όσοι θέλουν να μιλήσουν, μια και δεν είμαστε πολλοί, να το δηλώσουν για να εκπονήσουμε τον κατάλογο με τους αγορητές. Ο κύριος Κούκαν, Λινκεβιτσιούτα, Γιαζοβιέτσκα, Μαρτάν, Μαρτά. Όποιος άλλος παρακαλώ θέλει να μιλήσει, να το δηλώσει. Κύριε Κούκαν, έχετε το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτά που μας είπατε για τον αγώνα, λάθος τα είπατε. Όχι ένα, δύο μηδέν κερδίζουμε. Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Βάις ε, και το δεύτερο ο Χαμσίκερ. Ε, σας καλωσορίζουμε λοιπόν ε, κύριε Επίτροπε Κοιτάξτε, το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης απασχολεί πολλούς πολιτικούς ε, στην ε, Ένωση και πάρα πολλοί και στην ΑΦΕΤ και στην ΙΤΡΕ συζητούν ε, το θέμα των περιφερειακών συμφωνιών για την ενέργεια. Όλα αυτά ενέχουν και μία κοινωνική διάσταση. Και εσείς προηγουμένως είπατε ότι πρέπει να υπάρχει η κοινωνική διάσταση. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μας ενδιαφέρει το θέμα των κοινωνικών διακρίσεων λόγω ηλικία. Φέτος ε, έχουμε το έτος της Ενεργειακής Ένωσης και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον ε, στα πλαίσια αυτού ε, του έτους ε, θα ληφθούν μέτρα για ηλικιωμένους. Μιλάμε για ψηφιοποίηση και για άλλου είδου επιτεύγματα. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ελπίζω κύριε Επίτροπε να εργαστείτε με επιτυχία για τα θέματα αυτά μέχρι να υπάρξει τελική πρακτική εφαρμογή και τα ήθελα να σου ευχηθώ ε, κουράγιο από καρδιάς. Εγώ θα μιλήσω λιθουανικά και περιμένω μέχρι να βάλετε τα ακουστικά σας. Και εγώ, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που προσφέρεται να υπάρχει συνεργασία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Εσείς είστε ένας από τους πιο πεπειραμένους και είσαστε αρμόδιος ε, για ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι σημαντικός και από πολιτικής πλευράς. Προφανώς και αναφέρομαι στην Ενεργειακή Ένωση. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι η ενεργειακή πολιτική συνδέεται άμεσα με τις μεταφορές, ε, τη γεωργία, τη βιομηχανία και επίσης σωστά επισημάνατε ότι όλα αυτά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Είμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, και ένα πράγμα θέλω να επισημάνω. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ενεργειακή ένδυα. Εσείς ταξιδεύετε πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ έχω παρακολουθήσει πολλές συναντήσεις στη Λιθουανία. Ένα λοιπόν από τα θέματα που θίγονται σε αυτές τις συναντήσεις είναι ότι για μας δεν αρκούν τα εισοδήματά μας για να καλύπτουμε τα έξοδα θέρμανσης στα σπίτια μας. Άρα δηλαδή, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κατατετούν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς ακριβώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενεργειακής ένδυας. Μιλήσατε για ένα 10% ε, πολιτών στην Ευρώπη που έχουν δάνεια ε, λόγω δαπανών θέρμανσης. Πάνω από 12% των ανθρώπων ε, δεν μπορούν να διατηρήσουν μια ικανοποιητική σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι τους. Άρα δηλαδή πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς είσαστε επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας. Να πω λοιπόν το εξής. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δικαιοστάσιο. Ε, να μην αποκόπτονται νοικοκυριά από ενεργειακό δίκτυο. Εσείς τι πιστεύετε για ένα τέτοιο είδους δικαιοστάσιο. Και κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε εδώ στην Επιτροπή για το ελάχιστο εισόδημα και απευθύναμε τα αιτήματά μας στην Επιτροπή είπαμε ότι αν δεν μπορεί να διασφαλιστεί το ελάχιστο εισόδημα, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής ένδυας. Εσείς τι πιστεύετε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και κάτι άλλο. Μιλήσαμε για τα διαρθρωτικά αλλά και για άλλα ταμεία και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον προτίθεστε να καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το θέμα της ενεργειακής ένδυας. Αυτά είχα να σας ρωτήσω και σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιαζοβιέτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε γιατί μας μεταφέρατε τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα της Ενεργειακής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή η τρομοκρατία λαμβάνει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και μορφές. Επαναλαμβάνω, η τρομοκρατία λαμβάνει όλο και διαφορετικές εκφάνσεις και μορφές. Μερικές φορές μας ευνηδιάζει μάλιστα. Είμαστε εξασφαλισμένοι απέναντι σε τρομοκρατικές επιθέσεις ό,τι αφορά τις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις. Ποια είναι η στρατηγική που θα μας εξασφαλίσει και την ενεργειακή ασφάλεια. Υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή μας ασφάλεια και πώς αντιμετωπίζουμε πιθανά τρομοκρατικά χτυπήματα. Thank Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις και πάνω απ' όλα ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο για τις χαρμόσυνες ειδήσει που μου έδωσε και τις ακόμη πιο ευχάριστες που μου έδωσε ο κύριος Κούκαν. Θα ήθελα συντομία να απαντήσω σλοβακικά. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της ε, απασχόλησης ε, των εργαζομένων άνω της ηλικία των 50 ε, ετών, πράγματι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ, ως 50 πρόσφατα μάλιστα έγινα 50 χρονών, σας λέω ότι σφίζω από ενέργεια. Άρα δηλαδή πρέπει πράγματι να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους ε, και σε σχέση με την τεχνολογία. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα αλλάζουν, ε, αλλάζουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζουν οι ε, παραδοσιακές ε, βιομηχανικές δομές. Για όλες λοιπόν αυτές τις ε, περιοχές πρέπει πλέον να υπάρχει ένα νέο πρότυπο και να δώσουμε τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Τώρα, θεωρώ επίσης ότι πράγματι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για τη διαβίου μάθηση. Ε, για αυτούς τους ανθρώπους πάντα ε, πιο προχωρημένης ηλικία. Από την πρακτική γνωρίζουμε ότι δεν είναι χρήσιμες ε, όλες οι πρακτικές διαβίου μάθησης και όσον αφορά στους νέους υποψήφιους που αναζητούν νέες δεξιότητες θα πρέπει και αυτούς να τους βοηθήσουμε να τις αποκτήσουν. Άρα δηλαδή πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ε, και θέλω να σας πω ότι εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό, θα επικοινωνήσουμε με, τη, με τους αρμόδιους. Δυστυχώς δεν ναι, μιλώ λιθανικά, γι' αυτό θα πρέπει να πατήσω στα αγγλικά στην κυρία Βλυνκεβιτσούτε. Σε ό,τι αφορά το θέμα του πώς η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει όλες τις πτυχές ε, του οικονομικού μας βίου. Έχετε δίκιο, δεν επηρεάζεται μόνο η ενέργεια, αλλά και οι μεταφορές και η γεωργία από την ενεργειακή μετάβαση. Επηρεάζεται ο οικοδομικός κλάδος, ε, οι εξορυκτικές βιομηχανίες. Όλοι αυτοί οι τομείς θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες που απαιτούσαν στο παρελθόν. Σήμερα οι εργαζόμενοι χρειάζονται πολύ περισσότερες ε, δεξιότητες για ε, ε, τον ψηφιακό, κόσμο και σίγουρα οι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να αποτελούν τμήμα των νέων σχολικών προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ένδυα, καταρχήν ακόμη προσπαθούμε να βρούμε τον ορισμό του τι εστί ενεργειακή ένδυα. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και τελικά επιλέξαμε τρία κριτήρια με βάση τα οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει πρόβλημα ε, με την ενεργειακή κατανάλωση. Το, ένα ήταν η θέρμανση. Δεύτερον, οι λογαριασμοί. Καταφέρουν ε, οι άνθρωποι να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους ε, της ενέργειας. Και τρίτον, μήπως ζουν σε ανθυγιεινές με υγρασία, για παράδειγμα. Έτσι, με αυτά τα κριτήρια προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε ένα, μια κοινή προσέγγιση και ένα κοινό ορισμό της ενεργειακής ένδυας, να κάνουμε κοινή αξιολόγηση και να μπορέσουμε να εκπονήσουμε πιο κατάλληλα μέσα για να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, αποσύνδεση ε, από τον ηλεκτρισμό ή από τη θέρμανση να μην θερμαίνει το σπίτι του κάποιο ε, ή να κόβει το ηλεκτρικό. Ακόμη και στη Γερμανία έχουμε μεγάλο αριθμό οικογενειών που κόβουν το ηλεκτρικό ή κόβουν τη θέρμανσή του, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στην νέα αγορά ηλεκτρισμού να έχουμε ε, πτυχές καταναλωτή, εκδημοκρατισμού της διαχείρισης της ζήτησης και επίση όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την ετοιμότητα των κρατών μελών να ενστερνιστούν τις προτάσεις μας. Όταν κανείς έχει στεγαστικό δάνειο και αντιμετωπίζει πρόβλημα, φυσικά δεν χάνει μέσα στο σπίτι του. Η τράπεζα του προσφέρει κάποια μεταβατικά μέτρα, κάποιες συμβουλές, δεν του κατάσχει αμέσω, δεν του δημεύει αμέσω το σπίτι που έχει ενυπόθηκο δάνειο. Προσπαθεί να βοηθήσει τον οφειλέτη να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Και αυτό θα βοηθούσε πολύ κόσμο στην Ευρώπη. Αν υιοθετούσαμε δηλαδή αυτή την προσέγγιση, αυτούς τους μηχανισμούς πριν κόψουμε σε κάποιον το ρεύμα ή τη θέρμανση. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τις εθνικές νομοθεσίες. αν υπάρχουν μεταβατικέ διατάξεις, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα θέσουμε επιτάπητο για να μην ε, ανησυχούν οι συμπολίτε μας τι θα γίνει τον επόμενο χειμώνα. Και να μην έχουμε άλλε τέτοιε διακοπέ ούτε από την παροχή ηλεκτρισμού ούτε από την παροχή θερμότητας δεν έχετε όνομα, κυρία μου, δεν μπορώ και ούτως άλλως κάθεστε μακριά και αν έχετε δεν μπορώ να διαβάσω. Για έτσι κάνω, δεν κάνω λάθος, είναι το όνομά σας. Αν κατάφερα να το προφέρω και σωστά. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, το συζητήσαμε και στο παρελθόν και τώρα με τη νέα κατάσταση η συζήτηση επανέρχεται στο προσκήνιο και διευρύνεται όλα. Η προστασία κρίσιμων υποδομών είναι σημαντικό ζήτημα. Άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά το θέμα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών. Και στην Ευρώπη τα κράτη-μέλη μας ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο και αντιμετωπίζουν όλο και πιο σοβαρά αυτό το θέμα. Τώρα, Χρειαζόμαστε κάποιε κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ και ποια θα ήταν η βέλτιστη κοινή προσέγγιση για να προστατεύσουμε τι κρίσιμε υποδομέ μα. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση και η καλύτερη λύση για να έχουμε τον υψηλότερο βαθμό ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαφοροποίηση των προμηθευτών μας σε ενεργειακά προϊόντα ή η καλύτερη διασύνδεση των συστημάτων μας. Οπότε αν έχουμε ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένη περιφέρεια, σε συγκεκριμένη χώρα, χάρη στις τεχνικές δυνατότητες που έχουμε, στις τεχνολογίες και στα καλά ε, σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή στη λελεγγύη μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είχαμε προτείνει όταν συζητήσαμε την ασφάλεια ανεφοδιασμού φυσικού αερίου. Ζητήσαμε ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων εκτάκτου ανάγκη. Και αυτό θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και στην αγορά ηλεκτρισμού, ηλεκτρικού ρεύματο. ώστε να υπάρχει αλληλοβοήθεια στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματο σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω ότι έτσι θα εξασφαλίσουμε τα εχέγγυα ότι αν κάτι συμβεί σε μία περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπόλοιπες περιοχές θα είναι έτοιμες να βοηθήσουν και να καλύψουν την ενεργειακή, τον ενεργειακό ανεφοδιασμό απάσα πάσα περίπτωση. Ο κύριος Μαρτάν. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Διπρόεδρο. Ξέρετε ότι οι λέξεις ε, έχουν ε, σημασία Κυρίω όταν είναι και γραμμένε, μιλάτε για Ενεργειακή Ένωση και αυτό με ενοχλεί κάπω, γιατί ξέρετε, Ενεργειακή Ένωση αυτό σημαίνει ότι προβλέπουμε καθολικέ ε, λύσει και μεθόδου διακυβέρνηση και διαχείριση καθολικέ. Μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε απόλυτα τι επικυριαρχίε των κρατών μελών. Εγώ θα προτιμούσα να μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εξορθολογισμό της ενεργειακής καταναλώσης. Αυτό θα μας φόβιζε λιγότερο. Πέραν αυτών, όλα αυτά που μας εξηγήσατε μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Και νομίζω ότι, όπως είπατε, όλα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν αν υπάρχει το καρότο, το κίνητρο. Πάντα χρειάζονται ένα κίνητρο περίεργος πώς. Και αυτό το κίνητρο, λοιπόν, θα πρέπει να αφορά ε, όλες τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές κτλ είτε πρόκειται επίσης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους μικρομεσαίους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι μεγάλες επιχειρήσεις, ε, τους αυτοπασχολούμενους, ε, θα πρέπει πάντα φυσικά όταν υπάρχει ένα κίνητρο, ο κόσμος θα προσπαθήσει να το ακολουθήσει. Και έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουν τα έργα και από τη φωνή που θα ξεκινήσουν τα έργα θα υπάρχει δημιουργία θέσεων απασχόληση σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους πολύ απλά γιατί πρόκειται για μια κλιμακούμενη κατάσταση. Το καρότο θα οδηγήσει σε κίνητρο και άλλους ε, τομείς. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερο στα, λόγια σας είναι ότι μιλήσατε για συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των ερευνητών και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει το βασικό κινητήριο στοιχείο, τον κινητήριο παράγοντα. Έτσι θα βρούμε νέες μορφές ενέργειας και έτσι θα διαμορφωθούν με πραγματικό τρόπο αυτές οι ενέργειες. Οι ερευνητές μας, τουλάχιστον στην Γαλλία και παντού στην Ευρώπη, ε, έχουν περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους και όλα ε, μάλλον οι δαπάνε και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη είναι περιορισμένες και έτσι λοιπόν η έρευνα και η ανάπτυξη μετακινείται προς άλλες χώρες που έχουν τις επενδύσεις, όπως είχε πει και ο στρατηγός Ντεγκόλ Στη Γαλλία όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος βρίσκει τον ψάχνουν. Προφανώς ε, εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Επικράτεια γιατί στη ΣΥΠΑ, στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε πολλές άλλες χώρες βρίσκουν καλύτερες συνθήκες και έχουν ε, τα μέσα τα που χρειάζονται και σεβασμό μεταξύ άλλων, και κύρος. Να σας κάνω και μια ερώτηση, την οποία ενδεχομένω να μην περιμένετε, κυρία Αντιπρόεδρε. Τι θα γίνει με την ε, πυρηνική ενέργεια. Ποιο είναι το μέλλον που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια και τι προβλέπετε γενικότερα σε ό,τι αφορά αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε για την ενεργειακή ένδυα. Κύριε Αντιπρόεδρε, τι προτάσεις έχετε για τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κρίση όπως είναι η Ελλάδα. Είπατε ότι είχατε μία επικοδομητική συζήτηση με τους υπουργούς στο Συμβούλιο. Στην Ελλάδα τον επερχόμενο χειμώνα οι πολίτες θα πληρώνουν πιο ακριβά την ενέργεια με την αύξηση του ΦΠΑ στο 24% και την εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμασης με αυτό της κίνησης. Επιπλέον φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στα καύσιμα. Το αποτέλεσμα θα είναι χιλιάδες οικογενειών να μην έχουν πρόσβαση σε θέρμανση και θα καταφεύγουν σε τρόπους που είναι περισσότερο ρηπογόνοι όπως είναι η καύση ξυλίας. Επίσης θα έχουμε οικογένειες που δεν θα έχουν ούτε ηλεκτρικό γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Είστε αισιόδοξο για την πορεία της Ένωσης προς την κατεύθυνση αυτή. Εγώ πάλι δεν είμαι γιατί αυτά τα μέτρα επιβάλλονται στην Ελλάδα από τους δανειστές, οι οποίοι δεν είναι άλλοι παρά οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη δυστυχώς είναι μόνο στα λόγια και όχι στα έργα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και το λόγο έχετε εσείς για να απαντήσετε στις τελευταίες ερωτήσεις. να απαντήσετε και να συνοψίσετε. Προκειμένου να πάρουμε και ένα μήνυμα από την όλη συζήτηση. Uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε κύριε Μαρτών, πιστεύω ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι ένα project που δεν αφορά απαραίτητα στην μεταφορά της κυριαρχίας, αλλά πρόκειται για την συγκέντρωση σωστών ε, προσεγγίσεων που αφορούν στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Και είναι σαφές νομίζω ότι βλέποντας κάποιους τομείς όπως είναι η κλιματική αλλαγή και ανταποκρινόμαστε σε θέματα που έχουν σχέση με την ενεργία και ασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες και οι πιο πλούσιες χώρες στην Ευρώπη σίγουρα ε, βρίσκονται σε καλύτερη θέση εάν η συνεργασία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει υποστήριξη για το εγχείρημα αυτό της ε, Ενεργειακής Ένωσης και η υποστήριξη δεν είναι μόνο εδώ από τα γραφεία των Βρυξελών ε, πρέπει να σας πω ότι αυτό το εγχείρημα το έχω συζητήσει και με τους Υπουργούς ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Πήγα και στο ΝΑΤΟ για να παρουσιάσω αυτό το εγχείρημα ε, στους Υπουργούς Μεταφορών, στους Υπουργούς ε, Κοινωνικών Υποθέσεων. Ήμουνα στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι το συνέστημα που αποκτά κανείς είναι θετικό. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει υποστήριξη όλων αυτών στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό έχω ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συζήτησα με πολίτες και με στη Γαλλία και στη Γαλλία όπου εξεπλάγει για το πόσοι ήρθαν για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ε, Τέτσαν πολλές κρίσιμες ερωτήσεις, αλλά όχι παρατηρήσεις. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι στον τομέα αυτό μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα αν συνεργαστούμε και αν χρησιμοποιήσουμε τα ατού των κρατών μελών και αν η Ευρώπη μπορεί να αποδείξει ότι συνεργάζεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι αυτό το εγχείρημα επιβάλλει κάτι το ανεπιθύμητο σε επίπεδο κρατών μελών. Από την άλλη πλευρά ψάχνουμε να βρούμε πώς μπορούμε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε καλύτερα. Ε, ποιος είναι καλύτερος τρόπος για να γύρουμε γέφυρες στην Ευρώπη, έτσι ώστε η Ευρώπη στο σύνολό της να αποφεληθεί από τη συνεργασία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπάρχει ε, σωστή υποστήριξη του εγχειρήματο και στα τρία επίπεδα. Και χάρη στη Συμφωνία των Παρισίων έχουμε ένα πολύ καλό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν που συζητάμε εδώ και που προτείνουμε με τις νομοθετικές μας προτάσεις είναι να συσταθεί ένα σταθερό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θέλουμε βέβαια να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ε, για... Ε, προγράμματα ενεργειακά για να μπορούμε να δούμε πόσα και ποια κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλλουν, ε, πόσα αυτά τα εθνικά προγράμματα μπορούν να κουμπώσουν έτσι ώστε να έχουμε και αυτό το θετικό ε, μοσαϊκό ε, στην ευρωπαϊκή ενέργεια. Συνεργαζόμαστε πολύ συχνά με τα δίκτυα των ε, πόλεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διασφαλίσουμε ότι στο κατώτατο επίπεδο θα έχουμε την ίδια υποστήριξη και στενή συνεργασία. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία και όταν ταξίδευα στην Ευρώπη πρέπει να σας πω σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για αυτό το εγχείρημα. Γιατί το θέμα είναι τι θέλει κανεί να επιτύχει. Θέλει να επιτύχει μέσα από την καλή συνεργασία να υπάρχουν καλύτερε ενεργειακέ τιμέ. Να έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Ε, να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, με καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους και επίση να αναζητήσουμε λύσεις ε, έτσι ώστε να γίνεται και καλύτερη απορρόφηση των, ε, ε, των εφευρέσεων στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό για καινοτομίε ας πούμε στο Silicon Valley στην Αμερική, αλλά μπορώ να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Ε, πριν από δύο εβδομάδες που ήμουν στο Eindhoven, γιατί εκεί οργανώθηκαν από την Προεδρία διάφορες εκδηλώσεις, πρέπει να σας πω, να σας πω ότι εξεπλάγει θετικά, γιατί στο Eindhoven υπάρχουν ε, περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά 10.000 ανθρώπους από ότι στο Silicon Valley. Απίστευτο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό, ότι έχουμε ε, το δυναμικό των εφευρέσεων και στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η έννοια του ε, κόστους ωφέλους. Τώρα λοιπόν καταρτίζουμε και νέα στρατηγική έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αυτό το ε, νέο εργαλείο του επιμερισμού του κινδύνου, έτσι ώστε όλοι οι ερευνητέ να μπορέσουν να ξεπεράσουν την αρχική φάση και να φέρουν αυτά που ανακαλύπτουν στην αγορά. Ε, βέβαια, τελικά αποφασίζουν τα κράτη-μέλη, γιατί γνωρίζετε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ε, σαφείς κανόνες και αναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν μόνα τους για το ενεργειακό τους μείγμα. Εμείς επιμένουμε ότι δεν υπάρχει διαφωνία και από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να συνεχίσουν ή να ε, αναστείλουν τη χρήση της ε, πυρηνικής ενέργειας, αυτό γίνεται σε ανώτατο επίπεδο ασφάλειας όπου τηρούνται πλήρως ε, οι πιο αυστηρές προδιαγραφές. Νομίζω ότι επ' αυτού υπάρχει απόλυτη συνεννόηση και όλοι συνεργαζόμαστε. Η τελευταία ερώτηση από τον κύριο Φουντούλη αφορά στην κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρετε, εγώ έχω επισκεφτεί την Ελλάδα αρκετές φορές και νομίζω ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το αναγνωρίζουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αλλά και άλλων πολιτικών κομμάτων που τους έχω σταντήσει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες διότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να μετατραπεί σε ενεργειακό ε, κόμβο λόγω αυτού του νέου αγωγού που κατασκευάζεται από την Κεντρική Ασία προς την Ευρώπη και γι' αυτό αλλά και για τα πετρελοκοιτάσματα στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο γι' αυτά αλλά και γιατί ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό ηλιακής ενέργειας για όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η περιοχή πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αυτό θα ήταν προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών και οφείλω να σας πω ότι συμμεριζόμαστε πλήρως το αίσθημα που επικρατεί, αλλά επίσης ε, και το βάρος που φέρουν οι Έλληνες πολίτες για να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα που, ε, με τα οποία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη η χώρα. Εγώ πιστεύω μέσα από τη συνεργασία και τη σκληρή δουλειά των Ελλήνων αυτή η κατάσταση κρίση δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί. Αυτά. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ε, την παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Δείξατε κάποια θέματα ε, τα οποία η Κομισιόν πρέπει να τα σκεφτεί κυρίως το θέμα της ε, ενεργειακής ένδυας, αλλά και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την δίκαιη αντιμετώπιση εκείνων ε, που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σε επίπεδο ενέργειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς, αποκινούμε τα κράτη-μέλη, να προσφέρουμε ικανοποιητική χρηματοδότηση κυρίως για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όχι όμως μόνο για τους νέους, αλλά και για αυτούς που είναι άνω της ηλικίας των 50 ετών. Θέλουμε λοιπόν μία συνεχή αναβάθμιση του ε, ενεργού πληθυσμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Το 2016 είναι το ενεργειακό έτος ε, και όταν θα έχουν κατατεθεί όλες μας οι προτάσεις, ε, τότε ίσως μπορούμε να ξανασυναντηθούμε για να δούμε πώς κατορθώσαμε τελικά όλα αυτά που λέγονται να τα εντάξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί να συνεργαστούμε και κατά τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που με καλέσατε. Πρόεδρος, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και απαντήσετε σε τόσες ερωτήσεις. Το πρόγραμμά σας συνήθως επικεντρώνεται ε, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ήτρε περισσότερο. Εμείς είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και, και για μας το θέμα της ενεργειακής μετάβασης είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει μεγάλο δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και αφορά και τα κοινωνικά θέματα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Καλύψαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, την ενεργειακή ένδυα, τα ποσοστά ανεργίας και σας είμαστε ευγνώμονες για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Και είμαι βεβαία ότι θα μας ξανάρθετε σχετικά σύντομα. Ωραία, προχωράμε στο επόμενό μας θέμα. Αφορά την αξιοποίηση στο έπακρο του δυναμικού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντέμψκι. Παρακαλούμε κύριε εισηγητά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα πολωνικά. Θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση του έργου μας και των τροπολογιών, γιατί τις τροπολογίες εξετάζουμε. 358 τροπολογίες κατατέθηκαν επί του σχέδιου έκθεσης, κάτι που αποδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον των πολιτικών ομάδων για την έκθεση αυτή παρά ήταν ζωηρό θα έλεγα το ενδιαφέρον, μακάρι να ήταν λίγο ε, λιγότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις τροπολογίες τους ε, και να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους σκιώδης ηγητές. Είχαμε τέσσερις συναντήσεις μαζί τους και εργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά. Μέχρι στιγμής καταλήξαμε σε 23 συμβαστικές τροπολογίες, ε, για τις οποίες υπάρχει μέχρι στιγμής συνένεση και θα ήθελα στην επόμενη μας συνάντηση να συμφωνήσουμε και τα υπόλοιπα εκκρεμή θέματα και να διεκπαιρεώσουμε ή δυνατόν το θέμα των τροπολογιών. Είναι πραγματικά ανεκτήμητη για μένα η συνεργασία με τους συναδέλφους και τους σκιώδης ηγητές ιδιαίτερως. Πιστεύω ότι άσχετα με την πολιτική παράταξη στην οποία είναι και ο καθένα, όλοι συμφωνούμε για ορισμένα θέματα. Για παράδειγμα, να απελευθερώσουμε το δρόμο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, συμφωνούμε ως προς την αντιστοιχεία δεξιοτήτων και πραγματικών αναγκών της αγοράς. Ε, συμφωνούμε να αρθεί αυτή η αβεβαιότητα η κανονιστική και τα κανονιστικά εμπόδια ή ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιριών. Μερικές φορές, ενώ ο στόχος μας είναι κοινό, ε, μας ε, χωρίζουν οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούμε στην αποτύπωση των ιδεών μας. Γιατί από τη μια όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε καλές θέσεις εργασίας και άριστες ε, συνθήκες για τους ε, εργαζόμενους για να μπορέσουν να επιτελέσουν με ποιοτικό τρόπο την εργασία τους και να ε, αναπτυχθούν και ατομικά και υψηλές προδιαγραφές, αλλά αυτό έρχεται μερικές φορές σε αντίφαση με την αδύρυτη πραγματικότητα, γιατί η ζωή είναι δύσκολη και είναι δύσκολη πολλές φορές και η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μερικές φορές προσπαθούμε με μία διατύπωση να συμβιβάσουμε κάποιες αντιμαχόμενες έννοιες όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να είναι μεν ανταγωνιστικές και ταυτόχρονα να προστατεύουν ε, και να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους. Η κυρία Πρόεδρος το γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρούμε τη σωστή διατύπωση και να συνδυάσουμε μερικές φορές και αντιφατικούς στόχους. Και έχουμε και πολλές διμερείς πολλές φορές συζητήσεις για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες διατυπώσεις. Έχαμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, επί του σχεδίου έκθεσής μου Και εκεί ε, υπάρχουν σημαντικές απόψεις για τις ε, γεωγραφικές διαφορές, τις περιφερειακές διαφορές και την ανάγκη χρηματοδότηση μερικές φορές αυτών. Επίσης ε, και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών ήταν σημαντική. Εκεί αναφέρονται οι δραστηριότητες στις περιφέρειες που είναι πιο μειονεκτικές και δεν χρησιμοποιούν αρκετά τα κοινοτικά κονδύλια. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές των περιφερειών στο περιβάλλον που δημιουργούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η, την κεφαλαϊκή θέση που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τον κίνδυνο φερεγγιότητας τους. Θα πρέπει να περιορίσουμε αυτό το κίνδυνο αφαιρεγγιότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ίσως με κάποιες δράσεις της πολιτικής συνοχής. Αυτά εν ολίγης. Ευελπιστώ πάντως ότι θα καταφέρουμε στο εγγύς μέλλον να διεκπαιρεώσουμε τις εργασίες για τις συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστώ και πάλι τους συνεισηγητές και σκιώδησηγητές και ελπίζω ότι τον Ιούλιο θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας την έκθεση ώστε να καταφέρουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου να διεκπαιρεώσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τούν. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την διαδικασία που μας έχει εξηγήσει τώρα και τους υπόλοιπους όδους εισηγητές. Όντως, πολύ Έχουμε δείξει ενδιαφέρον για τα ευρύτερα θέματα και για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νομίζω ότι και οι εκφράσεις που διοργανώσαμε στι επιτροπέ μας έκαναν να σκεφτούμε σε ό,τι αφορά τις επαχθείς ε, και διπλές ρυθμίσεις, νομίζω διπλές. Ε. Αυτό ακούσαμε και αυτό τονίστηκε Καταλαβαίνουμε ασφαλώς ότι και η ρύθμιση ε, εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, δεν μπορεί να καταργηθεί, θα πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στη χρηματοδότηση, αλλά να δώσουμε και φορολογικά κίνητρα, προκειμένου δηλαδή να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες μέσω της φορολογίας. Προφανώς και όλος ο κλάδος των προσόντων, της εκπαίδευση, της απόκτησης νέων προσόντων είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες. Πριν από μια-δύο εβδομάδες είχαμε και την, ε, την ατζέντα για τις ψηφιακά, τα ψηφιακά προσόντα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι και αυτό, προκειμένου να έχουν οι εργαζόμενοι τα σχετικά και απαραίτητα προσόντα. Ένας άλλος κλάδος της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Κατανοούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν και περιλαμβάνονται στην έκθεση. Και ο εισηγητής επεσήμανε ότι υπάρχουν ε, πολλά γλωσσικά θέματα διατύπωσης και υπάρχουν διάφορες που εκφράζονται όλοι ε, μαθαίνουμε ένα από τον άλλον αλλά υπάρχει καλή θέληση και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σύντομα, ελπίζω μέχρι τον Ιούλιο, σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο και περιβάλλον στο οποίο μπορούν να ανθίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ πέρα λοιπόν ε, αυτός είναι ο αποτελέσμα σκοπός. Φυσικά σεβούμενοι πάντα τις αρχές της επικουρικότητας. Αλλά να δημιουργηθεί μια σωστή ατμόσφαιρα. Ε, ένα πλαίσιο όπου θα υπάρχει και αντίκτυπος και θα συνεχίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, όπως λέγεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λακή Πρόεδρος. Λόγο Περνάντες για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου ε, του Εμίλιαν Πάβελ, του σκιώδου συγγητού μα που δυστυχώς κολλείεται παρόλο που πολύ θα ήθελε να είναι παρόν και θα μεταφέρω τα σχόλιά του. Θα ήθελα καταρχήν εκ μέρους του σκιώδου συγητού να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας για την προσπάθεια που έκανε μέχρι τώρα και για την συνεργασία που επικράτησε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ήταν πολύ θετικές μέχρι τώρα οι Συζητήσει. οι Σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες έχουν καταθέσει πολλοί άριθμε τροπολογίε με στόχο να βελτιώσουν το κείμενο εξάρτητα τη σημασία που δίνει η ομάδα μα στις μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά προασπίζοντα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τη θέση του. Επίση, όπω αναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα αριθμιστικό ή κανονιστικό περιβάλλον ή πλαίσιο ε, πρόσφορο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα διευκολύνει τις επενδύσεις και θα αποτελεί εφαλτήριο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συμμετέχουν σε ένα κλάδο που καταφέρει και άντεξε σε μεγάλο βαθμό στην κρίση και θα αποτελέσουν ε, κλειδί για την ανάκτηση ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, γιατί τους άλλους δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα πρέπει να προσπίσουμε τους εργαζομένους, το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για τους μηχανισμούς ε, και για το κατά πόσο τα φορολογικά κίνητρα είναι τα πιο κατάλληλα μέσα για κάτι τέτοιο. Γιατί πολλές φορές τέτοιο είδους ε, κίνητρα αποβαίνουν εις βάρος των, του μισθολογικού κόστους και της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ε, θα ήθελαν να τονίσουν την σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων που θα αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγοράς, θα είναι επικαιροποιημένη και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα στους εργαζομένους μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σταθούμε και αυτό να επισημάνουμε την ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Και πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην κατάρτιση, στην επιμόρφωση και στις δεξιότητες, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Αυτή είναι η άποψη του σκιώδου συγγετού μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό, την ανάγκη να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό, δίκαιο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά που έχουμε. Μόνο έτσι θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, γιατί το χρειαζόμαστε και πιστεύω ότι για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στην Μαρτίνα Τζεμπάλαβα από την ομάδα του Άλτα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που κάνει. Και βλέπουμε ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο και χαίρομαι που έχουμε καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Και προς το παρόν ε, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν ξέρουμε φυσικά τι θα γίνει σε τελική ανάλυση. Πέρα από την πλάκα όμως χαίρομαι για τις συμβαστικές τροπολογίες που τονίζουν τέσσερα σημαντικά στοιχεία που με απασχολούν ιδιαίτερα. Καταρχάς, ε, μιλούν για την πρόθεση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το θέμα αυτό, γιατί το έχω αναφέρει πολλές φορές. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και η συμπεριφορά με επιχειρηματικό τρόπο. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε οι νέοι μας να είναι πιο αισιόδοξοι και να έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά το πώς τρέχουν η επιχείρηση και να δείχνουν πνεύμα επιχειρηματικότητας σε ό,τι κάνουν στη ζωή. Γι' αυτό μου αρέσει λοιπόν το Erasmus for Young Entrepreneurs για νέου επιχειρηματίε και πιστεύω ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να προωθούνται από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Δεύτερο στοιχείο, κάτι άλλο που μου αρέσει στι ε, τροπολογίε, στι συμβαστικέ, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τον ρόλο που παίζει για την αύξηση τη απασχολησιμότητας γιατί σε κάποιε περιπτώσει έχουμε υπερβολική επικέντρωση σε κάποια προσόντα που δεν βοηθούν. Τρίτο θέμα, όταν μιλάμε για ένα σταθερό περιβάλλον, όντω, όπω τονίζει ο εισήγητη, οι επιχειρήσει θέλουν νομική βεβαιότητα και ένα σταθερό περιβάλλον προκειμένου να μπορούν να ευδοκιμούν. Εκ παραλλήλου, και αυτό έχει προσθεθεί στι συμβαστικέ τροπολογίε, χρειάζεται στοχευμένα μέτρα οι μικρομεσαίες ε, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να προσλαμβάνουν ε, άτομα υψηλή ε, κατάρτισης. Άρα χρειαζόμαστε ένα σταθερό και υψηλή ποιότητα επίπεδο. Και τελευταίο θέμα. Να αναφερθεί η δυνατότητα περικοπής των εξόδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των νέων τεχνολογιών μέσω της ψηφιοποίησης, το e-government για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς αλλού για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Και θεωρώ ότι αυτά θα θα συζητήσουμε και στις ε, συνεδριάσεις των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σιλικιώτης, παρακαλώ. Πρόεδρε, αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον συνάδελφο Κραζοντεύσκη για την καλή συνεργασία και την όλη δουλειά που επιτελεί. Ε, με αφετηρία την τοποθέτηση που κάναμε στην πρώτη συζήτηση για την έκθεση για τι προοπτικέ απασχόληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταθέσαμε και εμεί ε, τροπολογίε επί του κειμένου. Είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που βλέπουμε πω η συνεργασία και με τι άλλε πολιτικέ ομάδε και κυρίω με τον εισηγητή είναι αγαστή και λαμβάνουν υπόψη και δικέ μα ευαισθησίε. Στα γενικά σχόλια που καταθέσαμε τροπολογίες για δημόσιες ε, επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, ε, εμείς θεωρούμε ότι είναι αγκές οι δημόσιες επενδύσεις για δημιουργία ανασφαλών και αξιοπροπών θέσεων εργασία, για κοινωνική ανάπτυξη, για προστασία των εργαζομένων και κυρίως για προστασία των συλλογικών του δικαιωμάτων. Επίσης τονίσαμε ε, και τον καταστροφικό ρόλο που έπαιξαν τα μέτρα, τα μνημονιακά μέτρα λειτουργούνται στην ανάπτυξη, ειδικότερα σε κάποιε περιοχέ τη Ένωση, οι οποίε οδήγησαν σε φτωχοποίηση των λαών, διαλύουν τα εργασιακά δικαιώματα και των κοινωνικών ιστών, αφού με τα μέτρα αυτά έπληξαν και τι ε, ε, συλλογικές ε, ε οδήγησαν και σε ιστορικά υψηλά ποσοστά συμπολιτών μα στην αργία, ιδιαίτερα ανάμεσα στου νέου. Ε, θεωρούμε ότι ε, είναι και σημαντικές οι τροπολογίες μας, ε, ειδικότερα στην, ως αυτές που αφορούν τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου Juncker. Βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές, εκείνες ειδικότερα που είναι σε ύφεση, δεν υλοποιούνται προγράμματα, γιατί ακριβώς η αρχιτεκτονική του σχεδίου Juncker είναι να έχουμε πρώτα ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς ρίσκο ε, και αυτό οδηγά πολλέ μεγάλε εταιρείε να μην επενδύουν σε αυτέ τι χώρε. Ε, και δείχνουν ότι οι χώρε όπως η Ελλάδα και η Κύπρο, που πλήγηκαν περισσότερο και με το χειρότερο τρόπο από τα μνημονιακά μέτρα λιτότητα, ε, δεν έλαβαν καθόλου επενδυτικά προγράμματα στο πρώτο εξάμεινο του 2016 από το πακέτο ούτε και ακόμα και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ενώ βλέπουμε ότι ελάχιστε επενδύσει έγιναν στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Τα πιο, κρατο, τα πιο πάνω κράτη-μέλη στον Νότο είναι αυτά που αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα νεανικής και γενικής ανεργίας, καλπάζουσα μετανάστευση των νέων, περικοπές μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων και βεβαίως ξύλωμα του κοινωνικού κράτους. Αντίθετα, βλέπουμε ότι χώρε όπω η Γερμανία άντλησαν τεράστια κονδύλια, κάτι που δείχνει ε, πω προφανώ όταν αφήνουμε την πρωτοβολία σε ιδιωτικά χέρια, τότε οι εταιρείε αυτέ χωρί να λαμβάνουν κανένα ρίσκο, να επενδύουν σε κράτη-μέλη με ήδη αθούσαν οικονομία και έχει σε περιοχέ που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι γι' αυτό που πιστεύουμε πρέπει να, να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη, δημόσιε επενδύσει, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίε είναι και η ε, σπορδιλική στήλη τη οικονομία τη Ευρώπη, ιδιαίτερα στι χώρε που έχουν μεγάλα ποσοστά ανεργία. Πέραν όμω των παρατηρήσεων μα αυτό, παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και θεωρούμε ότι ε, μέσα σε επικοδομητικό πλέμμα, στην επόμενη συνάντηση των σκιώδων ισογητών στις 28 του Ιούνιου, μπορούμε να βρούμε και άλλες συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ. κυρία Ζδάνοκα έχει το λόγο. Yes, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Σιγητά για την πολύ καλή σας δουλειά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τους σημασμούς που επιτεύχθηκαν στις ε, ε, συζητήσεις των σκιωδών. Κατατέθηκαν τροπολογίες που εστιάστηκαν κυρίως στην εκπροσώπηση των εργαζομένων και στον κοινωνικό διάλογο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στην έκθεση και βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για συνεταιρισμούς ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αυτές ε, από ό,τι ε, φάνηκε άντεξαν καλύτερα στην, στην κρίση και εκεί χάθηκαν λιγότερες ε, θέσεις απασχόλησης. Σε γενικές γραμμές είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με το πώς εξελίσσει η δουλειά. Ε, σκέφτομαι, ε, εύχομαι στον εισηγητή και στους υπόλοιπους ε, σκιώδες να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αντιλαμβάνεστε ότι είμαι σε πολύ δύσκολη θέση ε, που καλούμε να σχολιάσω αυτό το θέμα γιατί είχα αποκλειστεί από τη συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές που διοργάνωσε ο εισηγητής. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Κρασνοντέμσκι και ζητώ συγγνώμη αν πρόφερα λάθος το όνομά του, να τον ευχαριστήσω για το αξιόλογο έργο του και κυρίως για την ευφία του γιατί ο κύριος συζητητής είχε την κοινή λογική να αναγνωρίσει ότι οι τροπολογίες μας όχι μόνο ακολουθούσαν την γενική πορεία της έκθεσης, αλλά ήταν παρόμοιες με άλλες τροπολογίες. Και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που μου ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους έστειλα επιστολή στον πρόεδρο Έντελ και μου έδωσε κάποιες απαντήσεις που ήταν τελείως εκτός θέματος. Θα του ξαναστείλω λοιπόν επιστολή γιατί μιλά για το άρθρο 174.4 και για το άρθρο 209 που κατά τη γνώμη μου εξηγούν τη θέση των ομάδων ΕΛΚ, ε, ΓΚΟΕ και Σοσιαλιστών. Το 174.4 λέει ότι ε, εξαίρεση, με πρόταση του Προέδρου, οι τροπολογίε που κατατίθεται μετά την ε, ολοκλήρωση συζήτηση μπορούν να ψηφιστούν εφόσον πρόκειται για συμβιβαστικέ ή αν ανέκυψαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Τελείω άσχετο, εκτό θέματο η απάντηση του Πρόεδρου. Επίση, το άρθρο 209. Αυτό είναι ακόμη πιο αστείο. Λέει λοιπόν ότι τα άρθρα 14, 15, 16, 19, 38 48, 160, 162, 2 και 10, 165, 167, 169, 172, 174, αυτό που προανέφερα, το 176 παράγραφος 1, τα άρθρα 177, 178, 180, 182, λυπάμαι για τους διερμηνείς, περαστικά, 194 τα 197, 190 και 191 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών μουτά τη μουτάντης της συνεδριάς τη Επιτροπής. Αυτή ήταν η απάντηση που μου έδωσε ο πρόεδρος Έντελ. Τελείως ε, εκτός θέματος, άλλαν τάλλον. Και γι' αυτό θα ξαναστείλω επιστολή με τις ερωτήσεις μου. Και επίσης θα ήθελα να σας εκφράσω και να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη γιατί στη συντονιστική συνεδρίαση είχα την ιδέα να αγοράσω μία έκθεση για την Αλία, θεωρώντας ότι θα το αναλάμβανε ο αρμόδιος από την ομάδα. Δυστυχώς μου είπε ότι δεν είχε το χρόνο να ασχοληθεί με την έκθεση αυτή και ανακοίνωσε το θέμα στη γραμματεία μία εβδομάδα αργότερα. Δεν ήταν και τόσο αργά, ήταν προσωπική μου πρωτοβουλία, γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω στο σύνολο της Επιτροπής ε, την ταπεινή μου συγγνώμη. Αλλά και πάλι κατά κραυγή ξεσηκώθηκε. Και ότι μας είπαν ότι είναι ανυπόφορο, απαράδεκτο, ανίκιο, ανάρμοστο, έλλειψη σεβασμού. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη, συμπαθάτε με. Πώς όμως εξηγείτε ότι αποκλείσατε την ομάδα μου από τις συζητήσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες. Πώς χαρακτηρίζετε εσείς το γεγονός ότι δύο ομάδες, δηλαδή το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, συνέθλιψαν όλες τις υπόλοιπες ομάδες αγοράζοντας από κοινού μία έκθεση για τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους με τέσσερα μόρια χωρίς καμία συζήτηση και εκβιάζοντας οι υπόλοιπε ομάδες λέγοντας αν δεν μας αφήσετε να πάρουμε εμείς τι. Ε, ε, την έκθεση αυτή, στο μέλλον δεν θα σας αφήσουμε τίποτα. Δεν θα σας αφήσουμε καμία έκθεση. Αυτά δεν σας φαίνονται απαράδεκτα και ανυπόφορα. Δεν σας φαίνονται ανάρμοστα και ασεβή. Δεν σας φαίνεται αυτό σαν άρνηση της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Με σεβασμό προς τη δημοκρατία σας επέτρεψα να κάνετε όλα αυτά τα σχόλια τα οποία όμως δεν είναι αντικείμενο των όσων συζητάμε και των ε, θεμάτων που, επί των εργαζόμαστε για την έκθεση του εισηγητή. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και θα, θα συμμετάσχετε στη συζήτηση αυτή. Η συζήτηση την οποία ξεκινάται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των συντονιστών ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, δεν είμαι ενήμερη, δεν με ενημέρωσε κανείς και αυτό δεν είναι προβλέπωτο στην ημερήσια διάταξη. Σημειώσαμε τα σχόλια σας, ωστόσο. Για μια πραγματικά εντελώς διαφορετική έκθεση από αυτή που συζητάμε. Όπως είπε ο κ. Κρασναντεύσκη, η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόληση θα γίνει στις 13 και 14 Ιουλίου. Ελπίζουμε δε στην Ολομέλεια να περάσει τον Σεπτέμβριο. Ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο για να προσθέσει κάτι. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και σε άλλη προηγούμενη συνεδρίαση. Ίσως όμως επιθυμείτε να πάρετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Έχω την αίσθηση ότι με τα σχόλιά σας επιβεβαιώσατε κάτι που φάνηκε και στις συζητήσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες. Πολύ σπάνια στην πολιτική ε, υπάρχει τέτοια αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών παρατάξεων. Έχουμε αφενός την Άλντι, για παράδειγμα, που τονίζει την ανάγκη της επιχειρηματικότητας. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Φυσικά αναγνωρίζουμε την ανάγκη της επιχειρηματικότητας, άσχετα με την πολιτική ιδεολογία του καθενός. Και κάποιοι άλλοι επισημαίνουν τις κοινωνικές πτυχές. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Μάλιστα, εγώ είμαι ε, ναι με ένα αποσυντηρητικό κόμμα, αλλά με πολύ έντονο κοινωνικό προσανατολισμό, γιατί ξεκίνησε από τα συνδικάτα, από το Συνδικάτο Σολιντάρνος ε, για την Ελληνική. Οπότε μας ενδιαφέρει και η κοινωνική πτυχή, μας ενδιαφέρει ταυτόχρονα και η επιχειρηματικότητα. Οπότε από αυτή την άποψη όλα τα σχόλιά σας τα βρίσκω ενδιαφέροντα. Επίσης, θα ήθελα να πω στον συνάδελφο από την ΕΝΕΦ, τον κύριο Μαρτά, ότι εγώ είμαι κατά οποιοδήποτε αποκλεισμού και πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε αμοιβαίο σεβασμό στην κοινοβουλευτική μας εντολή, γιατί είμαστε εκπρόσωποι των ψηφοφόρων μας και αντιπροσωπεύουμε τις δικές τους απόψεις και αυτές μεταφέρουμε εδώ με το καλύτερο δυνατό τρόπο και αντίστοιχα και οι συνάδελφοι από τη Γαλλία αυτό κάνουν. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαίο σεβασμός μεταξύ μας στο όνομα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε. Πραγματι. Αλλά σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ε, απόσπαση των εργαζομένων, αυτό αποτελεί αντικείμενο τη πληροφορία του κ. Μαρτάν. Φυσικά και υπάρχει μάχη μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το ποιο θα κερδίσει το θέμα αυτό, την έκθεση αυτή. Και από όσο κατάλαβα, η ομάδα μας χρειάστηκε να δώσει πολλά ως αντάλλαγμα για να το πάρει και να το μοιραστεί με το ΕΛΚ. Δεν ήμουν παρούσα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά είμαστε... ανταγωνιζόμαστε στην ομάδα αυτή. Ανταγωνιζόμαστε παρά το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε, γιατί μας ενδιαφέρουν όλος ιδιαίτερος κάποιες από τις εκθέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απλά πρέπει να αποδεχτούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και στην παρούσα φάση έχουμε ένα πρόβλημα καθότι αναμένουμε για να συζητήσουμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα στη σημερινή ατζέντα, αλλά ε, ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Oettinger για τον αντεκτύπο της ψηφιακής ατζέντας. Θα καταφτάσει όμως τις 5.30 ο Επίτροπος. Η γραμματεία, τι συστήνει να κάνουμε. Μάλιστα. Ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε στις 5.30. Ελπίζω να επιστρέψετε. Ελπίζω γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερως. Πριν από μία εβδομάδα διοργανώθηκε ένα σεμινάριο για την ψηφιοποίηση και την ρομποτοποίηση. Ε, Υπήρχαν και κάποια μέλη της Επιτροπής στην Ακρόαση αυτή που συμμετείχαν και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα follow-up του σεμιναρίου της ημερίδας αυτής. Άρα, 5.30 θα ξαναξεκινήσουμε με τον Επίτροπο Oettinger ως προκεκλημένο μας. Διάλειμμα λοιπόν. Σας ευχαριστώ.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

Okay, friends, you can take your seat. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Έχει περάσει και η ώρα, αλλά με ιδιαίτερη χαρά έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Oettinger. Μας επισκέφθηκε και πριν καταφτάσετε εσεί. Συζητήσαμε θέματα Ενεργειακή Ένωση, Ενεργειακή Πολιτική και κατά πόσον αυτό επηρεάζει την αγορά εργασία. Εσείς δε είστε ακόμα πιο ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας ε, ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό σας και τα θέματα τα οποία εμπίπτουν και στην ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά την ε, απασχόληση και τις, ε, τα προσόντα. Χαιρόμαστε λοιπόν που σας έχουμε μαζί, μαζί σας μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Frau Vorsitzende, sehr Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και επίσης ε, σας ευχαριστώ πολύ για το ότι ως ε, Επιτροπή ενδιαφέρεστε για τα ε, ψηφιακά θέματα με τα οποία ασχολούμαι εγώ και μάλιστα τους τελευταίους μήνες θέσατε και πολύ εμπεριστατωμένες ερωτήσεις και στηρίξατε και τη δουλειά μας. Βλέπω επίσης ότι και η... έχετε και πολλές προσδοκίες όσον αφορά το αποτέλεσμα της δικής μας της δουλειάς. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι, ζούμε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης η οποία έχει ε, εκτενείς επιπτώσεις και θα έχει περισσότερο στο μέλλον σε όλες τις κοινωνίες. Έχουμε αφήσει πίσω μας ε, την επανάσταση, ε, την επανάσταση με την πρωτόλια έννοια, δηλαδή όσον αφορά το hardware, το software, τις τηλεπικοινωνίες. Σήμερα στην ψηφιακή εποχή βιώνουμε αλλαγές οι οποίες αφορούν τον τομέα, αυτό καθεαυτό, αλλά οι αλλαγές αυτές, και αυτό έχει σημασία, αφορούν περισσότερο τις ε, ψηφιακές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της ε, κοινωνίας. Παράδειγμα, ο κινηματογράφος, παντελώς ψηφιοποιημένος. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε σεναριογράφους, κοινογράφους, ε, ηθοποιούς, αλλά ακόμα και στους ε, θεατές εμάς. Άλλος τομέας, ο τομέας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπορείτε να ρωτήσετε ένα δημοσιογράφο. Η έννοια του είναι ο blogger και το δεύτερο δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση που υπήρχε παλιά, πότε κλείνει η αρχισυνταξία και πότε πάει το έγγραφο για να ε, τυπωθεί. Παλαιότερα υπήρχαν ε, Σαββατοκύριακα όπου την Κυριακή καθόντουσαν οι δημοσιογράφοι. Αυτά πια δεν ισχύουν. Τώρα online ενημερωνόμαστε για την πολιτική, την οικονομία, τα σκάνδαλα, τον αθλητισμό, τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτά για αυτά ενημερωνόμαστε ε, καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου και ως εκ τούτου ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση, αλλά αυτό βεβαίως σε κάποιο βαθμό εις βάρος της ποιότητας. Κινηματογράφος λοιπόν, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, τράπεζες, ασφάλειες, όλα αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί. Αυτοκίνητο βιομηχανία, η χρήση των αυτοκινήτων στην, ε, στις οδικές μεταφορές. Και εκεί υπάρχει διαδικασία της ψηφιοποίησης ή οι διανυκτερεύσεις, τα ξενοδοχεία, η πώληση σπιτιών, όλα αυτά ψηφιοποιούνται, οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω διαδικτύου και εμείς πιστεύουμε ότι το 90% όλων των μορφών παραγωγής και όλων των θέσεων εργασίας <clears throat> μετά από 5 μέχρι 15 χρόνια, το 90% λοιπόν θα έχει ψηφιοποιηθεί και αυτό καταλαβαίνετε θα συνεπάγεται πολύ σημαντικές αλλαγές για όλους τους εργαζόμενους. Στην πατρίδα μου, τη Γερμανία, μιλάμε για βιομηχανία 4.0. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε την τέταρτη επανάσταση στην οικονομία και στον χώρο της εργασίας, όμως ε, η βιομηχανία δεν ακολουθεί τον ίδιο διότι δεν πρόκειται μόνο για την παραγωγή, πρόκειται για τη μεταποίηση, για το εμπόριο, για υπηρεσίες ε, κάθε μορφής και πρόκειται και για τον κόσμο της εργασίας. Πρόκειται για την εργασία, την κοινωνία, όλα αυτά σε αυτό το ίδιο, με το ίδιο κριτήριο του 4.0. Άρα δηλαδή η Κομισιόν καλείται να καταδείξει τις δυνατότητες ε, που ε, θα οδηγήσουν στο να υπάρχουν λιγότεροι τιμένοι, να προκύψει ανάπτυξη, να προκύψουν θέσεις απασχόλησης. Και επίσης η Κομισιόν καλείται να προστατεύσει τους εργαζόμενους ε, και μέσα από την ψηφιακή εκπαίδευση και να τους μεταφέρει στον κόσμο της εργασίας ε, της επόμενης δεκαετίας. Στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας επικρατεί η ελεύθερη μετακίνηση. Εμείς προβλέπουμε ότι κατά τα επόμενα έτη κάθε χρόνο θα έχουμε περίπου 160.000 θέσεις απασχόλησης για εμπειρογνώμονες πληροφορικής επιπρόσθετα στις θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν ή ήδη ή, ή θα υπάρξουν. Αν λοιπόν δείτε το τι σημαίνει αυτό για τις επιπρόσθετες θέσεις εμπειρογνωμόνων ειδικών πληροφορικής και λάβετε υπόψη σας τις συνταξιοδοτήσεις θα καταλήξουμε στο ότι θα χρειαζόμαστε νέους ειδικού πληροφορικής ήδη από τους αποφύτους σχολείου ε, ε, φυσικούς, ειδικού ε, ειδικούς πληροφορικής, μαθηματικούς. Ε, από τις αναλύσεις λοιπόν που έχουμε κάνει, έχουμε καταλήξει στο ότι στα κράτη-μέλη και στις ε, περιφέρειες, ε, στα πανεπιστήμια μας, δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις φίτησης. Έτσι λοιπόν η δημιουργία ενός πανεπιστημίου δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου μόνο εφόσον υπάρχουν ε, αποτελεσματικές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, μπορούμε να προειδοποιήσουμε τα κράτη-μέλη για το ότι οφείλουν να προσφέρουν θέσεις φίτησης σε αυτούς τους τομείς και όχι μόνο να τις προσφέρουν τις θέσεις, αλλά και να τις χρηματοδοτήσουν. Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, εάν μία παραγγελία για ψηφιακές υπηρεσίες δεν παραμείνει στην Ευρώπη, αλλά πάει ας πούμε στη Νότια Κορέα, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι χάνουμε παραγγελίες γιατί στην Ευρώπη δεν μπορούν να εκτελεστούν και γιατί, γιατί δεν έχουμε αρκετούς ειδικού εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Κατά δεύτερον, Πέρα από τους ειδικού της πληροφορική, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας και του κόσμου της εργασίας, η ψηφιοποίηση αυτή σχεδόν για κάθε εργαζόμενο προϋποθέτει περαιτέρω εκπαίδευση στον χώρο της ψηφιακής πληροφορίας. Φεύγουμε από τον ανάλογο κόσμο και περνάμε στον ψηφιακό. Έτσι λοιπόν και ο ή οι εργαζόμενοι θα πρέπει και αυτοί να προχωρήσουν, να αλλάξουν ή οι εργαζόμενοι αυτοί θα δεχθούν περικοπή. Περικοπή στο μισθό τους. Κατόπιν τούτου, οι επαγγελματικές δεξιότητες η περαιτέρω μάθηση και εκπαίδευση. Είναι καθοριστική σημασία. Γι' αυτό το λόγο εγώ βρίσκομαι σε συζητήσεις με τα συνδικάτα και με τις ενώσεις εργοδοτών. Αυτή είναι η κοινωνική εταίρη. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει απαραίτητα ε, κάποια διαμάχη μεταξύ τους, κάτι άλλο. Ε, και οι δύο επιθυμούν την περαιτέρω εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όμως πρέπει να υπάρξουν πολλά περισσότερα. Αντίστροφα, εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και να τους πείσουμε να δεχθούν αυτή την προσφορά για το δικό τους το συμφέρον. Κατά τα άλλα, οι ψηφιακές ε, βασικές ε, γνώσεις και περαιτέρω εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, τους απλούς εργαζόμενους, αφορά και τον Γενικό Διευθυντή, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ε, τον Ελεύθερο Επαγγελματία, τον Επίτροπο. Αφορά η ψηφιακή ενημέρωση και γνώση ε, του CEO. Με λίγα λόγια, όλοι χρειαζόμαστε αυτές τις ψηφιακές γνώσεις. Όχι δηλαδή να μπορούμε όλοι να φτιάχνουμε λογισμικά ή εφαρμογές, εντάξει δεν λέμε αυτό, αλλά εκείνο που λέμε είναι να μπορεί κανείς να κατανοεί τα βασικά, το πώς μπορεί να αποθηκεύσει και να ανακαλέσει δεδομένα, ε, να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες, πώς προστατεύονται τα δεδομένα, τι σημαίνει ακριβώς ε, η General Data Protection Regulation, ο κανονισμός αυτός που αποφάσισε πριν από δύο μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυβερνοασφάλεια πώς μπορεί να ε, ενισχυθεί, ε, πώς ε, μπορεί κανείς να κλέψει δεδομένα, πώς μπορεί να αποφευθεί η βιομηχανική κατασκοπία, πώς μπορεί κανείς στο κινητό του τηλέφωνο να προστατεύσει τα δικά του τα προσωπικά δεδομένα και την προσωπική του ζωή. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι ο κάθε ένας από εμά έχει βασικές γνώσεις ψηφιακές γνώσεις και αυτά ισχύουν για όλους, ανεξάρτητα με το πιο ε, επαγγελματικό προφίλ έχουν. Γι' αυτό λοιπόν οι υπηρεσίες ειδικέ μου και εγώ χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ότι στο θεματολόγιο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες δεξιότητες, αυτό που αποφασίστηκε πριν από λίγες ημέρες, σε αυτό το θεματολόγιο προβάλλουμε το θέμα της ε, ψηφιακής παιδείας. Και όχι μόνο το προβάλλουμε, αλλά το αποδίδουμε και ιδιαίτερη σημασία. Αυτές, αυτά είναι και τα σχέδιά μας για το μέλλον. Όσον αφορά τώρα την ψηφιοποίηση, η ψηφιοποίηση στους ε, περισσότερους ε, τομείς αφορά το σύνολο της ε, αλυσίδας υπεραξίας. Από την αγορά προϊόντων μέχρι την αποθήκευσή τους, από την παραγωγή μέχρι την επαφή από μηχανή σε μηχανή, η επικοινωνία μεταξύ μηχανών M2M, B2B, C2C, ε, μέχρι να φτάσουμε στην παροχή υπηρεσιών ε, που αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται σε χή μέρος του κόσμου. Όλα αυτά λοιπόν από την στιγμή κατασκευής ενός αυτοκινήτου μέχρι την ε, παροχή υπηρεσία κινητικότητας επηρεάζεται όλη αυτή η αλυσίδα. Δηλαδή ό,τι μπορεί να ψηφιοποιηθεί, ψηφιοποιείται. Θα μπορούσε βέβαια κανείς εδώ να αντιπαραβάλει ότι εντάξει να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία όπου θα αναφέρεται απαγορεύονται δεδομένα. Να λέει αυτό. Και ότι τα δεδομένα είναι το πετρέλαιο της ψηφιακής οικονομίας. Ε, χωρίς δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει ψηφιακή οικονομία. Όμως, ξέρετε, δεν γίνεται αυτό. Ε, δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε την ψηφιακή επανάσταση. Ε, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ε, χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαίρονται πάρα πολύ για αυτό τον καινούριο κόσμο. Έτσι λοιπόν, τις ανησυχίες των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων μπορούμε να τις αμπλύνουμε ε, λαμβάνοντας υπόψη το τι πρέπει να υπάρχει στις κοινωνικές, στις εργασιακές συμβάσεις, στις συλλογικές συμβάσεις αν θέλετε. Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί επίσης από τα κράτη-μέλη. Και αυτό που έχει πει σημασία είναι πώς μπορούμε να επιτύχουμε η αλλαγή των θέσεων εργασίας να μην οδηγήσει σε επιδίνωση των εισοδημάτων και της κοινωνικής θέσης. Όχι κάθε, κάθε άλλο να υπάρξει βελτίωση της κοινωνικής θέσης μέσω της ανάπτυξης. Εδώ και κάποια χρόνια έχουμε μία, τον μεγάλο συνασπισμό ο οποίος έχει λάβει και συγκεκριμένα μέτρα σε 17 κράτη-μέλη. Τώρα αυτό θέλουμε να το επεκτείνουμε και να πούμε ότι θα είναι για συνασπισμό και για ψηφιακές ε, δεξιότητες ε, και θέσεις απασχόλησης. Ε, τα, την προσφορά περαιτέρω απασχόλησης θέλουμε να την υλοποιήσουμε μέσα από συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τον τριτογενή τομέα και ε, εμπορικούς άλλους θεσμούς. Για όλα αυτά, μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένους στόχους. Και παράλληλα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές. Εν ολίγης, έχοντας κατά νου τη δυναμική της ψηφιακής τεχνολογίας, αν δούμε λιγάκι το τι κάνουν οι Αμερικανοί μας ε, εταίροι και πώς εκμεταλλεύονται την ψηφιακή τους υπεροχή. Αν δούμε λιγάκι πώς οι Κινέζοι σε επίπεδο οικονομίας μιμούνται κατά γράμμα τους Αμερικανούς, αν τα δει κανείς όλα αυτά τρομοκρατείται. Εγώ όμως είμαι σίγουρος ότι η δημιουργικότητα των εργαζομένων μας αλλά και των επιχειρήσεών μας επαρκεί είναι ικανοποιητική γιατί αν τελικά φτάσουμε σε μια ψηφιακή εσωτερική αγορά, σε ψηφιακές προδιαγραφές και ψηφιακά πρότυπα για την εκπαίδευση και την περαιτέρω κατάρτιση και αν θέλουμε να ε, στηρίξουμε τις υποδομές μας έτσι ώστε ε, πλέον να μην υπάρχουν ε, επενδύσεις χωρίς θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να τονίσω γιατί ξέρετε ανησυχούμε για την περιφέρεια. Ανησυχούμε για το ότι η περιοχή όπου βρίσκεται ένας φοροτεχνικός ή ένας οδοντίατρος, στην περιοχή αυτή μπορεί να μην υπάρχει ψηφιακό σήμα. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν θα δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Θέσει απασχόληση θα δημιουργηθούν εκεί όπου είναι πλήρω ανεπτυγμένη η ευρυζωνικότητα. Άρα δηλαδή επενδύσει θα γίνονται σε νέα επαγγέλματα και σε νέες περιοχές και αυτό ε, μας οδηγεί στο να θεωρούμε ότι η ψηφιακή υποδομή είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάθε ε, μορφή ψηφιακής ε, διαίρεσης πρέπει να αποφευθεί και ψηφιακή διαίρεση της κοινωνίας τι σημαίνει μπορεί να υπάρξει μέσα από αυτούς που είναι ψηφιακοί γνώστες και ε, ψηφιακοί, ψηφιακά αναλφάβητοι ή περιοχές που είναι που έχουν ευρυζωνικότητα και άλλες που δεν έχουν. Εμείς με την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής όλα αυτά μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτά προβλέπει και το ε, σχέδιο Juncker. Εγώ μάλιστα κάνω σχέδια και για την περίοδο μετά το 2025. Να μπορούμε να προβλέψουμε και για τότε. Δηλαδή να προβλέψουμε για τις δυνατότητες, ικανότητες και για την ταχύτητα ε, ποιο θα είναι το δίκτυο, τόσο το σταθερό όσο και το κινητό κατά τα επόμενα έτη που θα είναι απαραίτητο για τη μεταφορά όλων των δεδομένων και για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης και στις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, σας ευχαριστούμε. Έχουμε ώρα για λίγες ερωτήσεις. Και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σφεν Σούλτς. Έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε Οτενιέρ. Θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας του έλκα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι βρίσκεστε μαζί μας σήμερα στην Επιτροπή και να συζητήσουμε το θέμα της ψηφιοποίησης της ε, οικονομίας και των επιχειρήσεων. Αυτό το θέμα, ξέρετε, μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν υπερνάει ούτε μια έκθεση ουσιαστικά στην ε, Επιτροπή που να μην αναφέρεται το ζήτημα. Και το θέμα της ψηφιοποίησης ε, επανέρχεται σχεδόν σε κάθε συζήτηση. Είναι λοιπόν ε, πολύ θετικό το γεγονό ότι βρίσκεστε εδώ να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Και η χρονική συγκυρία είναι πολύ ευτυχή. Στην προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, άλλωστε, συζητήσαμε το θέμα τη ατζέντα των νέων προσόντων, New Skills, με την Επιτρόπο Tyson. Και κοιτώντα ε, τι ε, παρεμβάσει, βλέπει κανεί ότι το θέμα τη ψηφιοποίηση διαρκώ ανακύπτει και στι 10 Ιουνίου η Επιτρόπο ε, παρουσίασε το New Skills Agenda. Όταν μιλάμε λοιπόν για New Skills, για νέα προσόντα, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και να μην αναφέρουμε το θέμα των ψηφιακών προσόντων. Αυτό για μας ως ΕΛΚ αποτελεί ένα από τα θέματα κλειδί. Όπως άλλωστε αποτελεί και ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας αποσχολήσουν για τον επόμενο καιρό στην Επιτροπή. Και πρέπει να πω, το έθιξαν και οι συνάδελφοι άλλωστε, διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει η χώρα η ψηφιοποίηση, θα πρέπει να την καθοδηγήσουμε και θα πρέπει ως Ευρώπη να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα αυτής, γιατί αλλάζει η εικόνα των επαγγελμάτων. Υπάρχουν όλο και πιο πολλά καινούργια ευρυδικά επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνουν και την ψηφιοποίηση και πολύ απλά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ψηφιοποίηση. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο, στους εργαζόμενους, την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να βιώσουν την ψηφιοποίηση, αλλά να τους δώσουμε και την δυνατότητα να δουν την ψηφιοποίηση όχι ως κίνδυνο, όχι ως ρίσκο, αλλά ως ευκαιρία. Γιατί συχνά συζητάμε για το κατά πόσο αποτελεί κίνδυνο, ρίσκο η ψηφιοποίηση. Λάθος πιστεύω την αυτή η συζήτηση δεν θα κλειστούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε ψηφιοποίηση. Δεν θα τεθεί τέτοιο θέμα. Υπάρχει και θα πρέπει να αποφεληθούμε από αυτήν, να εκμεταλλευτούμε. Αυτό ισχύει για όλους τους εταίρου, τους κοινωνικούς και λοιπού που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει διχασμός τη κοινωνία σε άτομα με ψηφιακά προσόντα και ψηφιακούς αναλφάβητους. Αυτό αποτελεί βασική έκκληση και αξίωση από, την πολιτική, από τους πολιτικούς και από τις επιχειρήσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να δείξω. Μιλήσατε για τη συνεργασία και με τα κλατη μελη Κάνετε συνομιλίες, αλλά αυτό που θα ήθελα να ακούσω είναι αν μπορούσατε να μας προσθέσετε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς ε, σκοπεύει η Επιτροπή Juncker να διεξαγάγει τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Γιατί στο θέμα της ψηφιοποίησης θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στην αντίληψη αλλά και στην υλοποίηση στα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, δεύτερο θέμα. Ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για τους ανθρώπους εκείνους που έχουν μειονεκτήματα σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση και τα ψηφιακά προσόντα. Η Επιτροπή Juncker και εσείς συγκεκριμένα πώς σκοπεύετε να προσεγγίσετε αυτούς τους ανθρώπους με τα προορισμένα ψηφιακά προσόντα. Πώς μπορείτε και πώς προτίθεστε να βοηθήσετε τα άτομα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, η Κιγιούτα Στάιρουκ. Ευχαριστώ κύριε Τιμέρ. Συμφωνώ με αυτό που αναφέρατε ότι αποτελεί ευκαιρία για μας η ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά, αλλά αυτό μόνο αν διαμορφωθούν με σωστό τρόπο οι συνθήκε και οι όροι πλαίσιο. Η έκθεση η οποία συνέταξα για την Επιτροπή Απασχόλησης ξέρω ότι την διαβάσατε επισταμένως και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή αντιμετώπισε το θέμα αυτό πιο πολύ από τεχνικής άποψης και ε, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο από την εκπαίδευση μέχρι την απασχόληση και ότι μόνο τότε θα πετύχουμε το στόχο μας. Και όντως αυτή την πρόκληση δεν μπορούμε να την ε, αντιμετωπίσουμε σε εθνικό επίπεδο, ούτε καν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο διεθνούς ανταγωνισμού. Πρόκειται για την πρώτη ύλη του μέλλοντος και οι ψηφιακές ικανότητες, τα ψηφιακά προσόντα αυτά θα πρέπει να καθοδηγηθούν και να προσανατολιστούν και στους νέους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επηρεάσει και τα κράτη-μέλη, γιατί είναι πολύ βασικό το ζήτημα της εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά τις ανατότητες σε σχολές κλπ. Αν χάσουμε την ευκαιρία και ίσως να έχουμε χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί μίλησατε για την Κίνα, για τις που έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά στην εκπαίδευση στον τομέα αυτό και είναι πολύ φιλόδοξες. Ό,τι αφορά την απασχόληση. Ένα από τα θέματα είναι η πιο ευέλικτη διαμόρφωση του ωραρίου εργασία, το οποίο θέλουν και πολλοί εργαζόμενοι. Αφετέρου, θα πρέπει να υπάρχει και μία ισορροπία στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Γιατί όντω θα υπάρχει ξεκοινωνικό αντίκτυπο αν είναι διαρκώ ε, προσβάσιμα τα άτομα αυτά. Και η ψηφιοποίηση, θα ήθελα να πω, ότι οδηγεί σε μεγάλο βαθμό σε επισφαλείς ε, θέσεις εργασίας. Πρόκειται για πολλούς αυτοαπασχαλούμενους οι οποίοι δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις κοινωνική προστασία και θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθούν τα σωστά κίνητρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί αν ξαφνικά βρεθούμε σε μια ψηφιακή αγορά όπου τα άτομα αυτά είναι το απασχολούμενα Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος χρήζει κοινωνικής βοήθειας. Γι' αυτό υπάρχουν και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν και ε, ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας τέταρτης γενιάς. Να προσαρμοστούν και οι αγορές εργασίας, ε, ε, η εξέλιξη των μισθών αν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτοαπασχολούμενων, τι ρύθμιση θα υπάρχει κρατική. Αυτά τα άτομα, οι αυτοαπασχολούμενοι, μπορούν να συνεννοηθούν για τις τιμές που θα χρεώνουν. Γιατί πρόκειται για πράγματα τα οποία στην παρούσα φάση τα συνεννοούνται τα συνδικάτα πέραν αυτού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να θεσμοποιήσουμε όλο και πιο πολύ την εκπαίδευση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί με, από την Βάντη, Βιτεμβέργη και έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις εκεί. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλου. τους, ε, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητα σε θέση να το πράξουν αυτό και θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους πόρους για να φροντίσουμε να μπορούν να το κάνουν αυτό και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους για το μέλλον. Από αυτό ξεπατεί το μέλλον μας για τις θεμελιώδεις, τις βασικές, αν θέλετε, ψηφιακές ε, ικανότητες. Συμφωνώ. Γιατί πέρα από την τεχνική γνώση χρειάζονται και τα κοινωνικά προσόντα. Το πώς θα αντιμετωπίζουν τα νέα μέσα, τη δημιουργικότητα, αλλά και ένα αυτόνομος τρόπος σκέψης. Μιλήσατε για τον τίποτα μέσα ενημέρωση όταν κανείς λαμβάνει ειδοποιήσει διαρκώς ανά πάσα ώρα και στιγμή και ξέρουμε πόσο εύκολα διανύμονται οι πληροφορίες αυτές πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά Αυτό θα απασχολήσει όλους τους μηχανικούς ε, λογισμικού και πολλά θα εξαρτηθούν άλλωστε και από την δημιουργικότητα στους άλλους τομείς. Άρα, πέρα από τις ε, τεχνικές γνώσεις, χρειάζονται και κοινωνικά προσόντα, θεωρώ. Αυτό από δικής μου πλευράς και δεν έχω ουσιαστικά ερωτήσει να σας απευθυνώ, απλά να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ, η κυρία Τσίμερ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπατε κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ο στόχος. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Θα το πω λιγάκι καθ' δηλαδή θέλουμε ένα κόσμο επιστημονικής φαντασίας, ένα νέο ψηφιακό κόσμο. Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να φτάσει κανείς εκεί. Και το θέμα είναι επίσης σε τι κόσμο ζούμε τώρα. Προηγουμένως είπατε ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για την απαραίτητη εκπαίδευση, δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις φίτηση, τα πανεπιστήμια δεν έχουν προσαρμοστεί. Αφού ισχύουν αυτά, τότε και εγώ διαρωτώ με το εξής. Στον ψηφιακό τομέα χρειαζόμαστε πάρα πολλές ε, θέσεις εκπαίδευσης. Από την άλλη όμως υπάρχουν άλλες πανεπιστημιακές σπουδές. Εγώ ας πούμε είδα ότι η Waterhouse PricewaterhouseCoopers λέει ότι μέχρι το 2030 θα καταστραφούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας στον τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας και της παραγωγής και ότι η ζήτηση μέχρι το 2030 θα περιοριστεί κατά 900.000 εργαζόμενους. Αυτό είναι οξύμορο. Από τη μια λέμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφιακά εκπαιδεμένοι, από την άλλη όμως ακούμε οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να περάσουν από το ένα τομέα στον άλλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να συνταξιοτηθούν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε νέα σχέδια που δεν θα αφορούν μόνο την εκπαίδευση των νέων που ξεκινάνε να σπουδάζουν, αλλά τι θα κάνουμε με αυτό το κοινωνικό δυναμικό που υπάρχει, που εργάζεται, που όμως θα κληθεί να αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικές προκλήσεις. Αυτές πρέπει να είναι διαδικασίες ε, οι οποίες θα έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει εδώ και πολύ καιρό αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πρόκληση. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο τώρα. Ήδη ελέγχθη ότι κυρίως ε, στον τομέα της περαιτέρω κατάρτισης γίνονται πάρα πολλές συστάσεις στα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει και χρηματοδότηση θέσεων για την περαιτέρω κατάρτιση. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν ε, μόνοι τους οι εργαζόμενοι, ε, δεν μπορούν ε, μόνοι τους να δουν πού θα βρουν θέση για να εκπαιδευτούν περαιτέρω ή να εκπαιδεύονται τα Σαββατοκύριακα, μα δεν γίνονται αυτά. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε τυχαία για το διασυνοριακό εμπόριο. Υπάρχει εδώ κίνδυνος ε, των ε, ε, επιχειρήσεων γραμματοκιβωτίου, των τελείως πλασματικών επιχειρήσεων. Υπάρχει και το θέμα της μετεγκατάστασης και το cloud working, το διασύνοριακό. Αυτά όλα είναι κίνδυνοι κατά την άποψή μου. Κάτι άλλο που θέλω να θέξω. Αυτές οι αλλαγές της κοινωνίας, αυτές οι αλλαγές, αν δει κανεί το σύνολο της αλυσίδας που δείξατε εσείς προηγουμένως, μα αυτές οι αλλαγές ε, δεν είναι μια ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε για το ωράριο εργασίας. Δηλαδή, ωράριο εργασίας το οποίο επειδή συνδέεται με την αυξημένη παραγωγικότητα θα πρέπει να περιοριστεί. Δηλαδή, να ξαναρχίσει η συζήτηση για το ότι ο περιορισμός του ορίου, ωραρίου εργασίας μπορεί να αποτελεί κίνητρο για εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις, βεβαίως να δίδεται η διασφάλιση σε αυτούς τους εργαζόμενους ότι και με μικρότερο ωράριο εργασίας θα μπορούν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Αυτά είναι θέματα που κατά την άποψή μου πρέπει να τα εξετάσετε. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να δώσουμε σε άλλους πέντε συναδέλφους να θέσουν ερωτήσεις τους, θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιδωλή στη χρήση του χρόνου, γιατί θα προλάβουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις του Επιτρόπου και δεν θα έχουμε και διερμηνία επαόριστο. Ίσως θα μπορούσατε να αρχίσετε τώρα με τις απαντήσεις και να δούμε αν θα προλάβουμε για δεύτερο κατάλογο. Αν θέλετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, παρακαλώ να είστε επιγραμματικοί. Η Τέρι, και... Ε, η ψηφιοποίηση δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο τους Γερμανούς, γι' αυτό θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ με κύριε Επίτροπε πολύ ενδιαφέρον που είπατε ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ε, ε, θα είναι ε, μέλη του ψηφιακού κόσμου και εγώ θεωρώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά και χαίρομαι ιδιαίτερος που το είπατε ξεκάθαρα στην ομιλία σας ότι το ψηφιακό θεματολόγιο δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία γιατί δεν είναι σαφές αυτό πάντα από την αρχή και θα επηρεάσει όλα τα Όλου του τομεί της κοινωνίας και την αγορά εργασία η ψηφιοποίηση, ακόμη και τον τρόπο λειτουργία της δημοκρατίας θα επηρεάσει. Θα καλύψει την κοινωνία σε όλες τις, πτυχέ πτυχές και εκφάνσει η ψηφιοποίηση δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Όπως είπαν οι συναδελφοί, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για μια συγκεκριμένη μορφή αυτού του ψηφιακού χάσματος, γιατί είπατε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αστικών και, υπέθ, και, αγρο, και αστικών περιοχών και υπαίθρου. Μόνο 9% των developers ήταν, ε, είναι γυναίκες, μόνο 19% εργαζομένων στον τομέα τεχνολογιών της πληροφορικής είναι γυναίκες και Πιστεύω ότι αν είχαμε συμμετοχή των γυναικών στον τομέα ε, πληροφορικής και τεχνολογιών θα είχαμε τεράστια κέρδη, γιατί μιλάμε για 9 δισεκατομμύρια ε, θα κερδίζαμε στα καθάριστα εθνικά προϊόντα με ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Η παιδεία είναι πολύ σημαντικό θέμα. Σε επιστήμες θετικές, ε, μηχανολογία, μαθηματικά και τεχνολογία έχουμε ελάχιστες γυναίκες πτυχίουχους. Θέλουμε επίσης πιο στοχευμένα προγράμματα και χρηματοδότησή της για να χειραφετήσουμε τις γυναίκες, να τις ενισχύσουμε και να γίνουν και αυτές επιχειρηματίες, να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή να συμμετέχουν περισσότερο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν αρκετές γυναίκες στο εργατικό δυναμικό τους. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρωτοστατήσει αυτό το θεματολόγιο έχετε τέτοιες προθέσεις για να κάνουμε πραγματικότητα την ισότητα των φύλων και στα θέματα της ψηφιοποίησης. Ο Ντομινίκ Μαχτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τεράστιο το θέμα, ευρύτατο. Ελάχιστο χρόνο μα έχει απομείνει, γι' αυτό και χαρίζω το δικό μου χρονογόρευση στον Επίτροπο. Ε, ε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και κύριε Τινιέρ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Tour αυτό που μας ε, καταδεικνύει τι ζούμε και τι βιώνουμε και τι θα βιώσουμε σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε μεταξύ δύο όλων. Εφορία από τη μία, ότι όλα θα πάνε καλά και τέλεια, και από την άλλη φόβος. Θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, η μέση οδός. Εμεί στην Επιτροπή Απασχόληση, λοιπόν, τι κάναμε. Μεταβήκαμε στο Silicon Valley. Την Amazon, την Facebook, την Google, την Intel και άλλε τέτοιε εταιρείε επισκεφθήκαμε. Και είδαμε πώς εργαζόντουσαν. Και το θέμα λοιπόν ήταν πώς μπορεί να προσαρμοστεί ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πάνω 50 εκατομμύρια Αμερικάνοι πλέον μπορούν να εργαστούν μόνο κατά ημιαπασχόληση. Δηλαδή, δεν υπάρχει απαραίτητα το ίδιο μοντέλο όπως αυτό που έχουμε στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά πλεονεκτήματα. Επισκεφθήκαμε επίσης το Πανεπιστήμιο του Μπερκλέη και μας είπαν οι καθηγητές «Αχ, ας είχαμε ένα τμήμα έστω και μόνο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου». Να προσέξουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και τα σχετικά μέτρα ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να διατυπώσουμε από κοινού τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να δώσουμε δυνατότητε μετεκπαίδευση, γιατί ήταν πολλού Ευρωπαίου οι οποίοι έχουν μεγάλη ζήτηση στη ΣΥΠΑ και μάλιστα κατεπηγόντω ακριβώ λόγω τη εκπαίδευσή του. Άρα, οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια έλλειψη οδηγεί και σε κάποια α, πλεονέκτημα. Και θα θέλαμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα όπως έχει και να έχουμε πραγματικά ουσιαστικά παραγωγικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως για την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε απόψε. Όντως, πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση αυτή που λαμβάνει η χώρα και προβληματίζει τους πολίτες. Έχουν πολλά ερωτηματικά γιατί έχουμε ε, πολλά στοιχεία της καινοτομίας που δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, πολλή ε, διασύνδεση και πολλές δεξιότητες που δεν ξέρουμε ακόμη τι μορφή θα πάρουν. Οπότε προβληματίζονται οι πολίτες ε, και φοβούνται μήπως υπάρξει μια πόλωση της απασχόλησης, κάτι που συνέβη και στις Ηνωμένε Πολιτείες με τέτοιες επιχειρήσεις ε, με πολύ ειδικευμένο προσωπικό, ευρηματικό, δημιουργικό και έχουν τα ζητούμενα προσόντα και από την άλλη έχουμε ε, ένα λιγότερο ειδικευμένο προσωπικό και ε, ανθρώπους που δεν έχουν ευκαιρίες απασχόλησης. Πώς θα διασφαλίσουμε και αυτές οι ενδιάμεσες απασχόλησης και αφετέρου θα ε, διευρύνουμε τις δεξιότητες των πιο ειδικευμένων. Είπατε, μιλήσατε για διασύνδεση, για αυτοματοποίηση. Πώς θα διασφαλίσουμε την ευρυζωνικότητα όχι μόνο στις αστικές αλλά και στις υπαίθριες περιοχές, στην Ήπεθρο περισσότερο. Δεν είμαι αφελής, είμαι κι εγώ ενθουσιώδης και πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση θα αποφέρει καρπούς, θα έχει πολλά πλεονεκτήματα και για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για τις περιοχές, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε και σε άλλα αγαθά, στην παιδεία, στην κατάρτιση ε, και για το αρχικό περιεχόμενο, να μην περιμένουμε το πανεπιστήμιο, να ξεκινήσουμε όπως και με την εκμάθηση γλωσσών από ε, προηγούμενο στάδιο της εκπαίδευσης ε, και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και επίσης σε διάφορες περιοχές να εμπλέξουμε και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτό συνέβη γιατί και οι ε, επιχειρήσεις ε, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης 4.0 είναι απαραίτητες, αλλά και η συνεργασία και η διασύνδεση με, τα, με τις διάφορες περιφέρειες. Με τι επενδύσεις ε, θα μπορούσαμε να ε, στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τις, τους περιφερειακούς φορείς για να προχωρήσουν σε αυτή την νέα εποχή. Κυρία Σόιντροβα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ λακωνική και θα υποβάλω απλώς τρία σχόλια και τρεις ερωτήσεις. Μιλήσατε για το θεματολόγιο των νέων δεξιοτήτων που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 7η Ιουνίου και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, με προβλημάτισε το γεγονός ότι οι νέες δεξιότητες θα πρέπει να ε, διδαχθούν από διδακτικό προσωπικό που έχει αυτές τις δεξιότητε ήδη και αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, αλλά πρώτα θα πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Αλλιώ ποιο θα διδάξει αυτές τις νέε δεξιότητε. Θα πρέπει πρώτα κάποιο να τις αποκτήσει για να τι μεταδώσει περαιτέρω. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη υποστήριξη των κρατών μελών. Επίσης, ε, ο συνδυασμός προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε, όπως η κατοίκον εργασία. Βέβαια, εδώ υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Η κυρία Σαντέρ μίλησε για κάτι παρεφερές. Είπε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις εταιρείες για να επιτρέψουν και εκείνες τις γυναίκες, στις μητέρες, στους γονείς να ε, δουλεύουν από το σπίτι χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές αυτές τεχνολογίες. Και επίσης, ε, οι ψηφιακές τεχνολογίες ε, δημιουργούν και ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και απειλές. Έγινε κάποιες έρευνες για τη χρήση των παιδιών που μπορούν να αγοράσουν από το ίντερνετ προϊόντα που θα ήταν πρόσθετα για αυτά. Και παιδιά κάτω το 16 μπορούν να αγοράσουν μέσω του διαδικτύου υνοπνευματόδη, ενώ δεν μπορούν να το κάνουν σε ένα μαγαζί, γιατί είναι ανήλικοι. Παρ' όλα αυτά, το διαδίκτυο τους επιτρέπει να αγοράσουν κάτι που κανονικά θα ήταν παράνομο. Οπότε προσοχή όταν στηρίζουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες, γιατί εμπεριέχουν και κάποιους κινδύνους πώς θα τα πλαισιώσουμε όλα αυτά και πώς θα αποσοβήσουμε αυτό το κίνδυνο κατάχρησης του διαδικτύου. Thank Uh, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια σχόλια λοιπόν και κάποιες ερωτήσεις και τώρα να ακούσουμε τον Επίτροπο Οεπτίνγκερ. Έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, Πολύ δείξατε το θέμα του σχολείου, του πανεπιστημίου, της εκπαίδευσης, ε, των σπουδών, ε, της περαιτέρω κατάρτισης ε, του εκπαιδευτικού προσωπικού και το θέμα των επαγγελματικών προσόντων. Εγώ είμαι φιλόδοξος, αλλά είμαι και ρεαλιστής. Δεν νομίζω λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα μου δώσουν κονδύλια για να εξοπλίσω τα σχολεία με υπολογιστές ε, ε, και προγράμματα υπολογιστών. Θα χρειαζόμασταν ε, πάρα πολλά κομπιούτερ, πολλούς φορητούς υπολογιστές, ανανέωση του λογισμικού. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Όμως, με 150 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο δεν μπορεί κανείς να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά. Το Σαββατοκύριακο, αν παρακαλέσετε τους πρωθυπουργούς σας να μου δίνουν 50 δις το χρόνο, κάτι θα κάνω. Όμως ε, όταν τα κράτη-μέλη λένε να περικοπεί ο ευρωπαϊκός προεπλογισμός στο Βερολίνο, λένε να δώσουμε περισσότερα ε, στη Γεωργία, στο Παρίσι λένε άλλα. Άλλοι πάλι λένε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν ε, θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές να γνωρίζουμε τι συζητιέται και σε τοπικό επίπεδο με δημάρχους, με τοπικούς βουλευτές, με φορολογούμενους. Με άλλα λόγια, εγώ δεν πιστεύω ότι οι βασικές αρμοδιότητες για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια ή για τον εξοπλισμό των ε, σχολείων και των πανεπιστήμιων ότι είναι δική μας ευρωπαϊκή υπόθεση. Δεν είναι. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Και αυτό το αναφέρω και στην έκθεση DC που είναι η ετήσια έκθεση για ε, το ψηφιακό δυναμικό των κρατών μελών. Ε, connectivity, υποδομές, θέσεις απασχόλησης, ερευνητικές επενδύσεις για την ψηφιακή τεχνολογία. Και κάθε χρόνο εμείς προκαλούμε ανταγωνισμό. Το γεγονός ότι είμαστε χειρότεροι στο θέμα των οπτικών ινών, ελπίζουμε να οδηγήσει το προλογούμενο σκεπτήμα γιατί να είμαστε τελευταίοι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι θα τεθεί το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες ε, θα πρέπει να είναι ένα σημαντικός παράγον των επόμενων εκθέσεων δέση, αυτών που ανέφερα προηγουμένως. Από κοινού με την ε, λουξεμβουργιανή. Προεδρία, πρέπει να σας πω, εγώ κάλεσα και τους 28 αρμόδιους υπουργούς για τις επιστήμες, για την παιδεία και αυτό σκοπεύω να το επαναλάβω και στο μέλλον και μάλιστα σκοπεύω ε, και να τους ε, ζητήσω να μου πούν συγκεκριμένα τι κάνουν ε, για να έχουν περισσότερες ψηφιακέ θέσεις στην εκπαίδευση, τι κάνουν στο επίπεδο της χρηματοδότησης για, να, για την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων ή το θέμα που έφυξε η κυρία Τσίμα. Δηλαδή, να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν ελεύθερο χρόνο από την εργασία τους για την περαιτέρω κατάρτισή τους. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα των κοινωνικών εταίρων. Στη Γερμανία είναι και θέμα περιφερειακής νομοθεσίας, σε άλλα κράτη εθνικής νομοθεσίας. Ε, στα πλαίσια όμως της best practice μπορεί κανείς να καταθέσει προτάσεις και εγώ να το κάνω αυτό. Τώρα, κατά πόσον αυτό θα το σεβαστούν οι κοινωνικοί εταίροι, καλό θα ήταν, αλλά ε, σε ορισμένα κρατημέλη κοινωνικοί εταίροι δεν συνεργάζονται, άρα δηλαδή εδώ καλείται ο νομοθέτης να επέμβει. Ετέθηκε το θέμα του διδακτικού προσωπικού. Ε, πολύ σωστά έχουμε 40, 50, 60 ετών δασκάλους ε, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και αυτούς πρέπει να τους καταρτήσουμε περαιτέρω. Όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο είχα μεγάλο σεβασμό για το δάσκαλό μου γιατί αυτός ήταν πολύ καλύτερος από εμένα. Σήμερα όμως ο δικός μου ο γιος ή οποιοδήποτε ε, στο θέμα ας πούμε της προπαίδειας είναι του είναι παντελώ αδιάφορο αν τα καταφέρνει καλύτερα ο δάσκαλο του ή όχι. Αυτό που τον νοιάζει το γιο μου είναι αν ο δάσκαλο είναι στο facebook και την Κυριακή το απόγευμα αν έχει πρόβλημα με τα μαθήματά του να μπαίνει στο facebook και ο δάσκαλο να τον βοηθάει. Ο δάσκαλο όμω πρώτον πρέπει να είναι στο facebook, δεύτερον πρέπει να έχει iphone και τρίτον βέβαια να μπορεί να απαντήσει σε αυτό που θέλει ο νέο. Εγώ ξέρετε είμαι ότι ότι οι μηχανές αναζήτησης μετά από λίγα χρόνια θα εντάσσονται, θα χρησιμοποιούνται ε, στις εξετάσεις. Εγώ όταν έκανα μπιτούρ, το απολυτήριό μου, μας επέτρεπαν να έχουμε το διαβήτη, ξέρω εγώ, το χάρηκα. Ε, ο πατέρας μου παλαιότερα δεν μπορούσε να έχει ούτε καν αυτό. Σήμερα όμως ε, έχουμε τα iPhone και αυτά επιτρέπονται στα, στις εξετάσεις που έχουν ε, τον ε, calculator ή ε, το Google, ας πούμε. Ποιος δεν χρησιμοποιεί το Google. Δεν υπάρχει ούτε βουλευτής, ούτε επιτρόπος, κανείς που να μην μπαίνει στο Google. Όμως, όταν τελικά το Google και οι μηχανές υπόλοιπες αναζήτησης θα μπουν μέσα στον εργασιακό μας χώρο, ε, δεν θα μπορούμε τότε να αποκλείουμε αυτές τις μηχανές αναζήτησης από τις εξετάσεις και από τα σχολεία. Άρα δηλαδή εδώ γίνεται λόγος και για την ε, ψηφιοποίηση ε, του διδακτικού, της διδακτέας ύλη και του διδακτικού προσωπικού. Και με τον τρόπο αυτό θα επανέλθει ο σεβασμός που θα νιώθουν τα παιδιά προς τους ε, δασκάλους τους, δηλαδή να μπορούν και οι δάσκαλοι στην καταμέτωπο εξέταση να είναι ε, καλύτερη από τα παιδιά σε θέματα ψηφιακών γνώσεων. Επίσης, εγώ σκοπεύω να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό κουπόνι. Αυτό θα ήθελα να υπάρχει. Ευρωπαϊκό κουπόνι για ποιους? Για όσους ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την περαιτέρω κατάρτισή τους. Ε, να έχουν τα κουπόνια, να παίρνουν και κάτι από το κράτος μέλος, ας πούμε άλλα 50 ευρώ και με αυτά τα κουπόνια να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάνε στα επιμελητήρια και οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ε, προσφέρουν εκπαίδευση για να αποκτήσουν αυτή την περαιτέρω κατάρτιση. Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό. Πρέπει λοιπόν, οφείλουμε τις ε, διατάξεις ε, των ε, συλλογικών συμβάσεων να τις εξετάζουμε και κάτω από το πρίσμα του κατά πόσον υπονομεύονται από την ψηφιακή τεχνολογία ή πώς πρέπει να μετατραπούν για να διατηρήσουν την ίδια αξία. Το πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει πλέον μια ευελιξία, ευελιξία στο χώρο, στο χρόνο. Το μειονέκτημα ποιο είναι ότι σήμερα ε, είναι κανείς ε, προσπελάσιμος όλο το 24ωρο και τα κλασικά ωράρια εργασίας. Και οι σταθερές θέσεις απασχόλησης με κοινωνικά επιδόματα για να υπάρχει κάποια εξασφάλιση για περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος, ε, γύρατος. Αυτά στον ψηφιακό κόσμο δεν θα είναι πλέον αυτονόητα. Υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα μειονεκτήματα. Παραδείγματο χάρη, αν ένα Σάββατο βράδυ έχει κριθεί ένα αθλητικό παγκόσμιο πρωτάθλημα ή γίνεται, ε, γίνεται διαγωνισμός τραγουδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την Κυριακή το πρωί όλα αυτά πρέπει να έχουν ήδη μεταδοθεί. Άρα δηλαδή δεν θα υπάρχει πια Σαββατοκύριακο. Ως εκ τούτου θα πρέπει κανείς να διερωτητή πώς μπορούν να θεσπιστούν κάποιες προδιαγραφές για να υπάρχει ποιότητα ζωής και πού μπορεί να υπάρχει κάποια ευολιξία, γιατί μόνο έτσι μπορούν να είναι και επιτυχημένες οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι στο θέμα των μέσων ενημέρωσης και στο θέμα της ε, ψηφιακής ε, εκπαίδευσης. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για τον, ε, για καταναλωτή. Δεν πρόκειται για τον εργοδότη, αλλά για τον εργαζόμενο, πώς ο εργαζόμενος μέσα σε αυτό τον καταιγισμό ε, πώς μπορεί και εκείνος ε, να διατηρήσει κάποιο επίπεδο ζωής. Παλαιότερα ε, διάβαζε κανείς εφημερίδες, διεθνή πολιτική, εθνική πολιτική, τα αθλητικά νέα, τις κηδείες, όλα αυτά. Σήμερα όμως αυτό δεν είναι εύκολο. Πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους να διαχωρίζουν να διαχωρίζουν την προσφερόμενη είδηση, τις προσφερόμενες εφημερίδες, τι είναι το YouTube, τι είναι οι εφημερίδες. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές ε, για, αυτήν, ε, για αυτόν τον ε, νέο ψηφιακό κόσμο. Και τελικά όταν μιλάμε για ποιότητα, για δημοκρατία, για ε, υποδάβληση μίσους για βία κατά των γυναικών. Ε, αν δεν θέλουμε όλα αυτά να τα δεχόμαστε, εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ποιότητα των ψηφιακών μέσων, αν δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα για τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, τότε με βάση τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε, θα πρέπει να προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον και online μπορούν να δοθούν απαντήσεις. Όταν διαβάζει κανείς την ε, εφημερίδα, εκεί ε, μπορεί κανείς να ελέγξει πολύ καλύτερα κατά πόσον ε, διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, κατά πόσον ενδεχομένω εξοραίζεται η βία κατά των ανθρώπων. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί κανείς να επιλέξει να διαβάσει όχι μια εφημερίδα. Όμως ε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεκδίονται αυτή της ευθύνη τους ε, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την τήρηση κάποιων προδιαγραφών. επίση ε, έγινε μια ερώτηση, αλλά η κυρία έφυγε. Διαπιστώνουμε, με βάση περιπτώσει, ότι ο αριθμός ε, των απασχολούμενων στον τομέα της πληροφορικής είναι τρομακτικά χαμηλός. Οι νέες γυναίκες ε, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στο Facebook δραστηριοποιούνται πάρα πολύ, αλλά δεν το έχουν κάνει επάγγελμά τους, οι φοιτητές της πληροφορικής, οι γυναίκες είναι πολύ λίγες. Και λίγες και στη φυσική και στην ε, ηλεκτρονική πληροφορία, πολύ λίγες γυναίκες. Ε, πρέπει λοιπόν στα σχολεία να ενθαρρύνουμε τις μαθήτριες ε, να επιλέγουν αυτούς τους κλάδους. Και αυτό μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχουμε το Startup Europe και εκεί προσπαθούμε στοχευμένα να ε, απευθυνόμαστε στις γυναίκες. Ε, εδώ έχουμε ως πρότυπο ε, την Αμερική, η Hewlett Packard και το Facebook. Αυτοί σε τακτά χρονικά διαστήματα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα μάλιστα, είχαν CEO γυναίκες. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα ότι οι γυναίκες ε, με τις κοινωνικές τους ικανότητες, την εργατικότητά τους ε, και την ε, ευφυΐα τους μπορούν να ανέβουν πολύ ψηλά στην σταδιοδρομία τους και με τον τρόπο αυτό να γίνουν πρότυπο για όλους όσους, όσοι θα ακολουθήσουν. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα που είχα να σας πω. Πολύ ευχαρίστω να επανέλθω μετά από ένα χρόνο για να μπορούμε να ξανασυζητήσουμε για την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί ή όχι και μην ξεχνάτε αυτό το Grand Coalition for Jobs and Skills. Ε, για μας λέξη ε, κλειδί είναι το να προσφέρονται περισσότερες ε, θέσεις ε, φίτησης στα πανεπιστήμια για, την, για τον κλάδο της πληροφορικής Υπάρχει το Business Europe, το Digital Europe. Θέλουμε να ακούσουμε από τους άμεσα εμπλεκόμενους που κρίνουν ότι πρέπει να παρέμβει ο νομοθέτης, να υπάρχουν θέσεις φίτησης και ε, έρευνας. Ε, ελπίζουμε μέχρι το τέλος ε, του έτους να έχουμε λάβει καλές αποφάσεις από τους κοινωνικούς τέρους. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επιτροπέ για την πολύ ε, ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, σύντομη και πολύ συναρπαστική και στην αίθουσα και στις συνεδριάσεις μας. Πάντα αισθανόμαστε ότι αυτό το θέμα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, γιατί μιλάμε για την ε, ανάπτυξη του νομικού μας, για την αγορά εργασία και συμπεριλαμβάνει και την κοινωνική ατζέντα, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση της κοινωνίας. Άρα, λέμε ναι στην προσφορά σας αυτή για να ξαναέλθετε σε ένα χρόνο περίπου. Ναι, θα βάλουμε και ημερομηνία, να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνάντηση αυτή και καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ. Hmm. down. <laughs>